So. Ladies and gentlemen. και κύριοι, ε, <clears throat> σας χαιρετώ στη σημερινή συνεδρίαση της, της Επιτροπής μας και αντίθετα με την παλιά μου μέθοδο αργήσαμε σήμερα αλλά ήθελα να παρίστανται όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι διότι θα προβούμε εις ε, την ε, συντακτική ε, Επιτροπή στη σύσταση σε σώμα. Η Επιτροπή αυτή διευρύνθηκε, τα νέα μέλη τα γνωρίζετε και έτσι δεν χρειάζεται να σας τα πω, θα το αποφύγω. Όσον αφορά τη δυνατότητα λήψεως αποφάσεως, ε, κανείς δεν την αμφισβητεί. Δηλαδή έχουμε απαρτία και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει web streaming για να μπορούν όλοι να συμμετέχουν. Ο στόχος είναι να μπορούν ε, καταρχήν να εκλέξουμε τον πρόεδρο και αντιπροέδρους και πρέπει να σας πω εάν μου πείτε να πω και μερικά λόγια πέραν της ημερησίας διατάξεως διότι εγώ θα ε, φύγω από την ε, θέση του Προέδρου σε αυτή την ε, συνεδρίαση. Δεν θα εγκαταλείψω όμως τη θέση μου χωρίς να έχω ευχαριστήσει θερμά όλους αυτούς οι οποίοι με βοήθησαν ή στο παρελθόν με καλή συνεργασία, επίπονη συνεργασία και το γεγονός ότι δεν συνεχίζω στη θέση αυτή δεν έχει καμία σχέση με το ότι δεν συμμετέχω και θα παραμείνω μέλος αυτή την εποχή θα θέλω να διαθέσω χρόνο αλλά έχω και άλλα να κάνω ε, θέλω να ευχαριστήσω όχι μόνο τους συναδέλφους αλλά και τους, ε, ε, τα μέλη της γραμματείας οι οποίοι δούλεψαν σκληρά σε αυτό το χρονικό διάστημα πολλές φορές κάποιος έφυγε από τη θέση του ο άλλος τον αντικατέστησε ευχαριστώ λοιπόν όλη τη γραμματεία διότι πολλές φορές μπορεί Δηλαδή, να σας δυσκόλεψα το έργο αλλά ελπίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν καλό. Θέλω να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους των διαφόρων πολιτικών ομάδων διότι συνεργάστηκα όχι μόνο με τους συνεργάτες από τη δικιά μας πολιτική ομάδα αλλά και από άλλες και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ε, σωστές και δίκαιες σχέσεις και ε, να ευχαριστήσω τους πάντες για την εξαιρετική εργασία στην Επιτροπή Βιομηχανίας η οποία είναι πολύ σημαντική επιτροπή για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οπότε πρέπει ίσως να ξαναπούμε πόσο σημαντική είναι η δουλειά την οποία κάνουμε και θέλω και πάλι να έχω πει τις ευχαριστίες μου. Και με αυτό Έρχομαι στο 5, δηλαδή το μόνο θέμα το οποίο θα διεκπαιρεώσω εγώ, δηλαδή την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων, ρωτώ το ΕΛΚ αν έχει μία πρόταση ε, για υποψηφιότητα και φαντάζομαι ότι η κυρία Ντελκαστήγιο θα θελήσει να κάνει μία πρόταση, γι' αυτό και της δίνω το λόγο. Κυρία Ντελκαστήγιο, έχετε το λόγο. Έρχομαι λίγο σε δύσκολη θέση, διότι η πρόταση που έχω να κάνω, ε, δεν ξέρω αν μπορεί να μου το επιβεβαιώσει και η γραμματεία, να με ενημερώσει η γραμματεία, γιατί δεν με ενημέρωσαν. Δεν έμαθα ποιον προτείνουμε. ναι, ναι, μπορώ βεβαίως, αλλά θα ήθελα να ξέρω ακριβώς πώς έχει διαδικασία και ο κανονισμός. Λοιπόν. Ακριβώς. Αλλά γι' αυτό και εγώ σκέφτηκα ότι πρέπει να κάνω μία πρόταση. Ναι, πρόταση για τον πρόεδρο, έτσι. Η κυρία Μάλια Σαρτόρη προτείνεται για πρόεδρο αυτής της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ωραία. Λοιπόν, είναι σαφής η πρόταση. Θα ήθελα να ξέρω αν η κυρία Σαρτόρη συμφωνεί με την ε, ε, υποψηφιότητα αυτή, δηλαδή αν είναι σύμφωνη να υποβάλει την υποψηφιότητά της. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, οπότε αν δεν υπάρχει άλλος ε, υποψήφιος θα ψηφίσουμε διαβοής. Ποιος είναι υπέρ της υποψηφιότητας της κυρίας Σαρτόρη. Εκλέξαμε την κυρία Σαρτόρη, καλή επιτυχία, συγχαρητήρια, όλες τις ευχές της Επιτροπής και παρακαλώ να αναλάβετε τη θέση εδώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για την υποστήριξή σας, διότι πέραν του γεγονότος ότι όπως γνωρίζουμε όλοι υπάρχει κάποια συμφωνία που αφορά όλες τις επιτροπές, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν γέννη, θα ήθελα παρόλα αυτά να σας ευχαριστήσω για τη θετική ψήφο που μου δώσατε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον προκάτοχό μου, τον πρόεδρο Ρόιλ, που όπως και εσείς ε, μπόρεσα να γνωρίσω πολύ καλά σε αυτά τα δυόμιση χρόνια και στη διάρκεια των ετών αυτών προείδρευσε με μεγάλη ικανότητα και ευφυΐα ε, της Επιτροπής. Εύχομαι να μπορέσω να σταθώ στο ύψος του και να μπορέσω όπως και αυτός να αγγιηθώ ότι θα γίνουν χρήσιμες, σωστές και θετικές εργασίες ε, ε, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία ε, είτε επιβεβαιώθηκαν, αλλά φυσικά και τα νέα μέλη που είναι πλέον ε, στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Να σας ευχαριστήσω και για τα όσα κάνατε στο παρελθόν και για τα όσα έκανε η Γραμματεία. Ε, εγώ παρακολουθούσα τις εργασίες ε, ως ε, μέλος ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω σήμερα και την Γραμματεία για το όσα θα εγγυηθεί στην Προεδρία και σε όλους εσάς για τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Ξέρω ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη η στήριξη των αντιπροέδρων, τους οποίους θα εκλέξουμε και θα προτείνουμε τώρα. Θα ήθελα μόνο να ρωτήσω αν πρέπει να προτείνω εγώ τα ονόματα ή ε, θα προτείνουν οι πολιτικές ομάδες. Ωραία λοιπόν. Για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποια πρόταση. κυρία Μαντουρέλ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ καταρχάς ε, να σας ε, ευχηθώ συγχαρητήρια ως νέα πρόεδρος και Εύχομαι να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Εγώ είχα συνεργαστεί και με την κυρία Σαρτόρη και σε άλλη επιτροπή στην προηγούμενη θητεία, στην Επιτροπή ε, Γυναικών και σα διαβεβαιώ ότι ήταν πολύ καρποφόρα και πολύ ευχάριστη συνεργασία. Συγχαρητήρια λοιπόν κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω αφού μου δώσετε το λόγο και τον πρώην Πρόεδρο για όλα τα όσα έκανα, τον κύριο Ρόιλ. Χέρμπερτ δεν ξέρω που είσαι αλλά ήταν τιμή και χαρά να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και σε ευχαριστώ διότι πάντα ήσουν ιδιαίτερα ανοιχτός και έτοιμος να διαπραγματευτείς και εργαστήκαμε με σκληρά αλλά πάντα σε καλό κλίμα και αυτό έπεφερε καρπούς εδώ στην Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθειά σου στη διάρκεια όλου αυτού του διαστήματος. Και τώρα να απαντήσω στην ερώτηση της Προέδρου. Η πολιτική μας ομάδα παρουσιάζει ως ε, πρώτη αντιπρόεδρο, την κυρία Πατρίτσια Τόγια και κατόπιν για τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Δημήτριο Δρούτσα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και την ε, πρώην Αντιπρόεδρο, την κυρία Άννη Ποδηματά, η οποία φεύγει από την Επιτροπή, αλλά θα ήθελα να την ευχαριστήσω για όλα όσα έκανε και για την αφοσίωσή της. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Grazie. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για τις ευχαριστίες προς τον κύριο Ρόιλ και τις, και τις συμβουλές προς εμένα. Έχουμε λοιπόν την υποψηφιότητα για την πρώτη αντιπροεδρία, την κυρία Πατρίτσια Τόια. Η υποψήφια δέχεται την υποψηφιότητα. Ναι. τα καταφατικά. Ευχαριστώ την κυρία Τόγια. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου. Αν όχι, προτείνω λοιπόν και πάλι να ψηφίσουμε διαβοής. Ε, συμφωνούν όλοι. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ λοιπόν. Καλό τώρα την κυρία Τόια ως πρώτη αντιπρόεδρο να έρθει εδώ στο βήμα. Περνάμε τώρα στη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου. Για τη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου υπάρχουν προτάσεις. Η κυρία Χολ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ επί τη εκλογή σας σαν πρόεδρο και να σας πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ όπως και τον κύριο Ρόιλ ε, διότι ήταν πάρα πολύ δίκαιος ε, ως ε, προείδρευε επί δυόμιση χρόνια την Επιτροπή αυτή. Θα ήθελα τώρα να ονομάσω εν ονόματι των φιλελευθέρων τον κύριο Γιάννη Ρόντερ, ο οποίος δυστυχώς δεν παρίσταται σήμερα αλλά θα ήθελα ήθελα να προτείνω το όνομά του για τη δεύτερη αντιπροεδρία. Ευχαριστώ πολύ για την υποψηφιότητα. Είμασταν ενήμεροι για την υποψηφιότητα και έχουμε λάβει και από τον κύριο Ρόντ γραπτός ε, την ε, αιτιολόγησή του για την σημερινή του απουσία αλλά και το γεγονός ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Ροντ δέχεται Υπάρχουν άλλες ε, υποψηφιότητες για τη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου. Κανένας άλλος, ωραία. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν προτείνουμε να γίνει εκλογή διαβοής. Συμφωνούμε όλοι. Bene. Καλώς, ευχαριστώ. Θα δούμε αύριο τον κύριο Ροντ εδώ στη συνεδρία τη Επιτροπής. Και τώρα για τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου έχει ήδη γίνει πρόταση για τον κύριο Δρούτσα. Δέχεστε την υποψηφιότητα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή σας. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι για την θέση του τρίτου αντιπρόεδρου. Κανείς άλλος. Ωραία. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν προτείνω να ε, κάνουμε την εκλογή διαβοή. Συμφωνούν όλοι. Ευχαριστούμε λοιπόν και καλό τον κύριο Δρούτσα να έρθει εδώ στο Προεδρείο. Και για τη θέση του τέταρτου αντιπροέδρου υπάρχει μια πρόταση ο κύριος Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας συγχαρώ επί τη εκλογή σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στη θέση αυτή. Έχω πείρα των δυσχεριών και είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει και θα περάσετε καλά διότι ε, όλοι οι συνάδελφοι είναι πολύ προσιλωμένοι ιδίω ε, αυτή την περίοδο. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Ρόιλ για την εξαιρετική και διεξαγωγή της Προεδρίας στο, στα πρώτα δυόμιση χρόνια να τον ε, συγχαρώ για την ανάληψη των νέων ευθυνών του και να προτείνω σαν τέταρτο αντιπρόεδρο τον ε, κύριο Τοζανόφσκι, τον ε, εκπρόσωπό μας, τον εκπρόσωπο της πολιτικής μας ομάδος. Χωρίς μικρόφωνο η πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Τσίτσιστερ. Κύριε Τοζινόσκι, δέχεστε. Ωραία, ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιο άλλο ο οποίο θέτει υποψηφιότητα για τη θέση αυτή. Όχι, ωραία λοιπόν και σε αυτή την τελευταία απορρίπτωση ε, ζητάμε εκλογή διαβοή. Αν συμφωνείτε. Ευχαριστώ πολύ. Έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Δελκαστήγιο. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αφού λοιπόν έχουμε πλέον πρόεδρο και τέσσερις αντιπροέδρους από τις πολιτικές ομάδες, θα ήθελα να διαβιβάσω και στους τέσσερις αντιπροέδρους και φυσικά την αποδοχή μου, την οποία την κάναμε με διαβοή, αλλά θα ήθελα να ευχηθώ συγχαρητήρια εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδος και να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο και να σας πω ότι μπορείτε να βασίζεστε στην υποστήριξη μας ε, και επιτρέψτε μου εδώ τώρα πριν ε, ολοκληρωθεί η σύσταση σε σώμα εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας θα ήθελα να εκφράσω πόσα πολλά οφείλει η ομάδα στον ε, απερχόμενο πρόεδρο που πραγματικά θεωρούμε ότι είχε μια άψογη προεδρία, ε, χρειάστηκε να εξισορροπήσει τα συμφέροντα όλων των πολιτικών ομάδων με την αμεροληψία την οποία πρέπει να διαθέτει ένας πρόεδρος. Κατά την άποψή μας αποτέλεσε υπόδειγμα και γι' αυτό και εγώ εξ ονόματος της ομάδας μου θα ήθελα να το επισημάνω δεδομένου ότι μόλις έγινε η αλλαγή της Προεδρίας. Ε, τίποτα άλλο, σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να χειροκροτήσουμε για άλλη μια φορά τον κύριο Ρόιλ. Καλώς. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το τμήμα της σύστασης σώμα της συνεδρίασης και μπορούμε πλέον να ξεκινήσουμε με τις συνήθεις εργασίες της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας. Στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης έχουμε την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Όπως γνωρίζετε, ε, έχετε την ημερήσια διάταξη στους φακέλους σας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο αίτημα. Υπάρχει αίτημα αντιστροφής των σημείων 3 και 15. Συμφωνούν οι εισηγητές. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν κάποιος ο οποίος να έχει κάποια αντίρρηση ή να κάτι άλλο επιπλέον στην ημερήσια διάταξη, μπορούμε με την αλλαγή αυτή να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Τα σημεία 3 με 15 αλλάζουν θέση. Συμφωνείτε όλοι? Ωραία. Δεν υπάρχει κανένας αντίθετος. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο σημείο 2. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Να σας πω λοιπόν ότι Επειδή υπάρχουν πάρα πολλέ ε, συνεδριάσει στη διάρκεια αυτή τη εβδομάδα, δεν θα είναι δυστυχώ διαθέσιμη διερμηνία σε όλε τι γλώσσε. Οι γλώσσε οι οποίε δεν είναι διαθέσιμε είναι τα εσθονικά, τα φιλανδικά, τα λετονικά, τα σλοβακικά και τα σλοβενικά. Αυτά λοιπόν από πλευρά μου για το γλωσσικό καθεστώς αυτή την εβδομάδα. Να περάσουμε τώρα λοιπόν στο σημείο υπαριθμών 3, το οποίο είναι το πρώην σημείο 15. Ενεργό συνεργασία με τους εταίρους πέρα από τα σύνορά μας στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής. Ζητώ συγγνώμη, σβήνω αμέσως το τηλεφωνό μου, είχα ξεχάσει να κλείσω το τηλέφωνο. Ε, με εταίρους πέρα από τα σύνορά μας λοιπόν μας, μια στρατηγική προσέγγιση για έναν ασφαλή, αηφόρο και ανταγωνιστικό ενεργειακό εφοδιασμό. Θα ήθελα να δώσω λοιπόν το λόγο στην Ντίτ Χέρτσχοκ. Α, συγγνώμη, η κυρία Χέρτσοκ δεν είναι εδώ. Η κυρία Μαντουρέλ λοιπόν θα λάβει το λόγο εξ ονόματός της. Συγγνώμη, η κυρία... Η κυρία Μέρκης. Επειδή η συνάδελφός μου δεν μπορεί να είναι παρούσα, μου ζήτησε να ε, διαβάσω το σημείο, την, ε, το σημείο σε σχέση με την εξωτερική πολιτική ενέργειας και θα το κάνω. Θα ήθελα ορισμένε παρατηρήσει να τονίσω σε σχέση με την έκθεση εκ μέρου ε, του εισηγητή. Καταρχά, ε, μία πλήρω ε, ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά ενέργεια είναι ένα σημαντικό τμήμα για μια επιτυχημένη εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το αντίστροφο ισχύει. Η ισχύ που προκύπτει από αυτή την ολοκλήρωση πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρω με το συνδυασμό τη τεχνογνωσία και των ικανοτήτων των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Τρίτον, η ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεξαρτησία της λήψης αποφάσεων σε άλλους τομείς ε, και, μόνο η αλληλεγγύη και ε, η συνεργασία των κρατών μελών μπορεί να εξισορροπήσουν αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να γίνουν συζητήσει σε σχέση με τι προκλήσει που αντιμετωπίζει στον τομέα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίσημε και ανεπίσημε συνεδριάσει των κρατών μελών σε επίπεδο υπουργών ε, με ε, την ε, με, με τους αντίστοιχους ε, επιτρόπους ώστε ε, να εξασφαλιστεί ολόκληρη ο εμφοδιασμός ενεργειακός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει επίσης να δοθεί μια διαπραγματευτική εντολή ώστε όλα, όλοι, όλοι οι τομείς που έχουν αντίκτυπο στην ενεργειακή πολιτική να ε, αντιμετωπιστούν αμέσως. Όλα τα σχετικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με, ε, τα, ενεργειακά προβλήματα, ε, με τα ενεργειακά προγράμματα που αφορούν και τρίτες χώρες πρέπει επίσης να είναι πάντοτε διαθέσιμα. όλα τα στοιχεία και όλες οι πηγές που έχουμε για τα στοιχεία πρέπει να τα να τα χρησιμοποιήσουμε ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δίωδος ε, μέσω για παράδειγμα του νότιου ή του βόρειου ε, διαδρόμου. Ε, επίσης πρέπει να συνεργαστούμε με την Αυστραλία, τον Καναδά, την Κεντρική Ασία και πολλές άλλες χώρες για την ενεργειακή πολιτική. Όσον αφορά τώρα τα ολοκληρωμένα as well as infrastructure. Τα δίκτυα παραγωγής ενέργειας ε, πρέπει επίσης να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να τα εξελίξουμε. Για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να πω ότι ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει την, την ανάγκη ύπαρξης ενεργειακών χαρτών, ε, όχι μόνο σε σχέση με εταίρους όπως η Ρωσία, αλλά και με εταίρους που έχουν κοινέ αξίες όπως ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και με σκοπό τις ανανεώσιμες, τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ε, ε, τη χρήση παλαιών αλλά και πιο συμβατικών μορφών παραγωγής ενέργειας, όπως επίσης και της πυρηνικής ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για τη συζήτηση αυτή έχουμε στη διάθεσή μας τρία τέταρτα. Υπάρχει ήδη ένας κατάλογος συναδέλφων με τους κοιόδης εισηγητές φυσικά συμπεριλαμβανόμενος. Κυρία Καλβάλιο, καταρχής. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς ε, να συγχαρώ και εσάς ε, και τους αντιπροέδρους, ε, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στη δουλειά σας για το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής θητείας. Ως και εισηγήτρια του ΕΛΚ θα ήθελα να συγχαρώ καταρχάς την εισηγήτρια για την δουλειά της. Πρόκειται για μια δουλειά η οποία είναι πραγματικά πολύ ισορροπημένη και θα ήθελα να τονίσω τα στοιχεία τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά στην έκθεσή της. Θα ήθελα επίσης να τονίσω δύο-τρία σημεία που θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να τα βελτιώσουμε περαιτέρω. Όσον αφορά τις ε, θετικές πτυχές της ε, έκθεσης. Ε, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απολύτως με τις προτεραιότητες ύπαρξης μιας εξωτερικής πτυχής της της αγοράς ενέργειας. Προσπαθώ να κλείσω το τηλέφωνο μου, αλλά δεν τα καταφέρνω.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 Λοιπόν, η βελτίωση της πρόσβασης στην αηφόρο ανάπτυξη για τις αναπτυσσόμενες χώρες και η ενίσχυση της ενεργειακής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από τα σύνορά της. Πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να έχει μία ενιαία φωνή θα δώσει πολύ μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στα διεθνή φόρα. Αυτό λοιπόν... Ε, αναφέρεται, όλα αυτά αναφέρονται ορθότατα στην έκθεση και συμφωνώ απολύτως. Όμως υπάρχουν τρία σημεία τα οποία θα ήθελα να τονίσω λίγο παραπάνω. Πρώτον, Έχει συζητηθεί το θέμα στο πλαίσιο της ε, πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Ανατολάς, προς Νότο ε, και προς Βορράν. Ε. Επίσης, νομίζω ότι η πολιτική Η ενεργειακή πολιτική είναι κάτι το οποίο λοιπόν πρέπει να μας ε, ε, απασχολήσει ιδιαίτερα. Ε, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα έπρεπε να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια. Θα έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη δημιουργία υποδομών στον τομέα των ενεργειακών. Ε, θα ήθελα λοιπόν να τονιστεί ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη έκθεση ε, η σχέση με την Νότιο Αμερική, με τον Νότιο Ατλαντικό, όπως επίσης και με τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, για να συμπεριληφθούν στις σχέσεις μας με τις χώρες αυτές ο τομέας της, η τομής της ενεργειακής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για το τηλέφωνο. Ο κύριος Τούρμες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ε, σας συγχαίρω και σας και τους αντιπρόεδρους για την ανάληψη των καθηκόντων σας και θα ξεκινήσω με έναν έκδοτο. Πριν από τρία-τέσσερα χρόνια ήμουνα στην ε, αντιπροσωπεία σχέσεων ΕΟΚ ε, Κίνας. Πήγαμε λοιπόν στην Κίνα, επισκεφθήκαμε διάφορους υπευθύνους και ε, αντελήφθηκα ότι δεν υπάρχει ενεργειακή πολιτική μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Υπάρχει μεταξύ της Κίνας και της Δανίας, της Γαλλίας και της ε, ε, Κίνας, της Γερμανίας και της Κίνας, αλλά τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα. Δηλαδή, η δανέζικη συνεργασία για την ενέργεια με ε, την Κίνα είχε μεγαλύτερο προϋπολογισμό από ότι αυτή της Ευρωπαϊκής Ενώσης για να καταλάβετε πόσο καλά οργανωμένοι ήμασταν. Και μάλιστα διαπιστώσαμε ότι για λόγους βιομηχανικής πολιτικής οι περισσότερες χώρες προσπαθούσαν να μην ανακοινώσουν τι κάνουν και αν υπήρχε, ίσως υπήρχε ε, μία εθνική ε, επιταγή να γίνει κάτι τέτοιο, όχι όμως ε, ευρωπαϊκή. Οπότε αν θέλουμε όντως να προχωρήσουμε όπου τα κράτη-μέλη και η ενεργειακή πολιτική και τα γεωπολιτικά συμφέροντα να καλύπτονται σε γενικό επίπεδο, θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και όπως αναφέρθηκε στον τομέα της συναπόφασης θα χρειαζόμαστε περισσότερες διμερείς συμφωνίες ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επίσης βασιζόμαστε για εξωευρωπαϊκούς προμηθευτές ε, για την προμήθεια ουρανίου, ενεργείας, ε, ενεργειακών πόρων Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ε, και να επιβάλλουμε ένα διεθνές νομικό καθεστώς διότι με το πετρέλαιο που έχουμε όλο και λιγότερες χώρες οι οποίες προσφέρουν περισσότερη ποσότητα τότε ε, βλέπουμε ότι Υπάρχει μεγαλύτερο μέρος της προμηθείας που δεν βασίζεται σε κανόνες αλλά στα παζάρια. Χρειάζεται λοιπόν ένα, ε, νόμι, ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να διέπει τις ανταλλαγές αυτές και στα πλαίσια του ΠΟΕ όταν μιλάμε ε, για, ε, ενέργεια για το εμπόριο ενεργείας θα πρέπει επίσης να ισχύει το ίδιο σύστημα. Ε, για άλλους τομείς πολιτικής όπως κλιματολογική πολιτική όπως και ένα άλλο θέμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι εάν οι εισαγωγές του Καναδά που έχουν διπλάσιες, τριπλάσιες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος από ότι ε, οι χώρες που καίνε πετρέλαιο, εάν ε, αυτό είναι καλό. Πρέπει να είμαστε δηλαδή συνεπείς και να πρεσβεύουμε ε, τις ίδιες αρχές προς όλες τις κατευθύνσεις. Και τέλος, όταν δείτε το χάρτη πορείας της ενεργείας στην Ευρώπη, στις Ηνωμένε Πολιτείε, στην Ιαπωνία, στην Κίνα, βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι τρία θέματα. Ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες ε, πηγές ενεργείας και ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν αυτές είναι οι μεγαλύτερες δυνατότητες των εξαγωγικών αγορών, οπότε θα χρειαστεί να καταρτήσουμε μία σχετική στρατηγική. Να βοηθήσουμε τις, ε, ε, τις κυβερνήσεις να καταρτήσουν συστήματα συγκεκριμένα όπως τις οικολογικές, τον οικολογικό σχεδιασμό αλλά και τα ε, έξυπνα δίκτυα και πρέπει να αναρωτηθούμε αν εμείς θα το πράξουμε ή αν θα αφήσουμε σε άλλες περιοχές του κόσμου όπως η Κίνα να κάνουν και να αναλάβουν αυτό το έργο για να δούμε τι μπορεί να γίνει ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου πολλές φορές φορές είναι οι τεχνολογικοί ε, ηγέτες, πώς μπορούμε δηλαδή ε, μπορούμε να συνεργαστούμε και να βοηθήσουμε τις αναδιόμενες ε, ενεργειακές αγορές. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Διούλ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την Πρόεδρο και να σας ευχηθώ καλή δουλειά για την επόμενη περίοδο. Επιπλέον θα ήθελα να συγχαρώ το συντάκτη της εκθέσεως διότι είμαι πεπισμένος όπως και οι προλαλήσαντες ε, ότι είναι μια πολύ ισοσκυλισμένη έκθεση όπου όλα τα θέματα τονίζονται σωστά. Το βασικό στοιχείο αυτής της εκθέσεως με την οποία συμφωνώ πλήρως είναι ότι χρησιμοποιούμε μία περίπλοκη προσέγγιση όταν εξετάζουμε τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες και ένα από τα βασικά στοιχεία αυτής ε, ε, της ε, ιδιομορφίας μπορεί να επιληθεί μόνο με την επίτευξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς. Δεν πρέπει λοιπόν να συγχαίουμε τα πράγματα. Από τη μία πλευρά να έχουμε δηλαδή μια εσωτερική ανταγωνιστική αγορά και διαφορετικές σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Έχω όμως να κάνω σχόλια ως προς τους συναδέλφους μας και εταίρους μας διότι είμαι βέβαιος ότι το κείμενο παρουσιάζει σωστά την κατάσταση, δηλαδή την κατάσταση των κρατών μελών όσον αφορά την εξάρτησή τους από τη Ρωσία που διαφέρει από τη μια χώρα στην άλλη και αυτό δεν αναφέρεται μόνο στην εισαγωγή του φυσικού αερίου αλλά και από το ισοζύγιο πληρωμών της ενδιαφερόμενης χώρας. Υπάρχουν δηλαδή ορισμένες χώρες οι οποίες εξάγουν, ε, ε, εισάγουν μεν λιγότερο αέριο αλλά εξαρτώνται πολύ περισσότερο από αυτό ε, από ότι παραδείγματο χάρη χώρες που ίσως ε, εξαρτώνται και 100% γι' αυτό και δεν είναι προφανές ότι μπορεί να υπάρξει αλληλεγγύη, αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών ένα άλλο θέμα ε, είναι η Κίνα το οποίο προανέφερε ένα συνάδελφος η Κίνα δεν τονίζεται αρκετά σε αυτή την έκθεση παρόλο που όλοι συμφωνούμε ότι από τις της πλευράς της καταπολέμησης της, ε, του, του φαινομένου του θερμοκηπίου θα πρέπει <clears throat> να υπάρξουν περισσότερες προσπάθειες και στην εταιρική αυτή σχέση θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο συγκεκριμένους τομείς. Τέλος θέλω να αναφερθώ ε, στις διάφορες πηγές ενεργείας ιδίως όσον αφορά το πετρέλαιο διότι πιστεύω ότι η εξάρτηση της Ευρώπης μας ε, υποχρεώνει ε, να ξεχνάμε την εξάρτηση από το πετρέλαιο παρόλο που υπάρχουν ανησυχητικά γεγονότα στην την Ιγυρία υπάρχουν τα αντίπεινα προς το Ιράν και οι κυρώσεις οπότε πρέπει να εξετάσουμε το θέμα του πετρελαίου και όσον αφορά γενικώ την ενέργεια, το ηλεκτρικά δίκτυα και το φυσικό αέριο πρέπει να τα αναπτύξουμε αλλά το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν διαχωρίζει μεταξύ του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου και πρέπει να δούμε αν εμείς μπορούμε να διατυπώσουμε προτάσεις για συγκεκριμένες στρατηγικές σε αυτό το χώρο. Τέλος θα ήθελα να μιλήσω για το χρονοδιάγραμμα. Είναι ατυχές ότι δεν γνωρίζουμε ε, ποιες είναι οι προθεσμίες για τα έγγραφα του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς λοιπόν μπορούμε να προσπαθήσουμε να καταρτήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει έκθεση Collins και αυτές οι δύο εκθέσεις που είναι αυτές που αντεστράφησαν Ίσως η έκθεση που εξετάζουμε είναι πιο σημαντική, αλλά εμείς πρέπει να ασχοληθούμε και με το χρονοδιάγραμμα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Δελκαστήγιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω και πολλά περισσότερα να προσθέσω από στα όσα ακούσαμε. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει να δούμε την έκθεση αυτή από κοινού με όλη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση αυτή δεν ε, θα γινόταν κατανοητή για τους ε, στόχους της ε, μεμονωμένα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις ε, διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών. Είναι κάτι βέβαια το οποίο είναι ξεχωριστό και θα το συζητήσουμε σε άλλη χρονική στιγμή, αλλά είναι αποφασιστική σημασία όταν προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας και σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Ένωση συγγνώμη, να μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω θετικά την παράγραφο υπαριθμών 8 που ζητά το Συμβούλιο να δίνει εντολές διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ε, υπάρχει ένα σημαντικό πρόγραμμα υποδομής ε, στρατηγικής σημασίας που επηρεάζει ε, την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της, ώστε να μην αναφερόμαστε μόνο σε διακυβερνητικά συμφέροντα, τα οποία θα μπορούσαν φυσικά να επηρεάσουν και τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω και την παράγραφο 11, όπου η συγγήτρια κατά την άποψή μας καταλήλως επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η αλληλεξάρτηση και η αλληλεγγύη ως ε, εργαλεία για να μπορέσουμε να ε, δούμε τι γίνεται με την ε, εξωτερική εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορυκτά καύσιμα και νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο αλλά ισχύει και για τον άνθρακα και θα πρέπει η αλληλεγγύη ε, να θυμόμαστε ότι δεν είναι δυνατή εάν δεν υπάρχει και διασύνδεση ε, την οποία αναφέρουμε πολύ συχνά εδώ, αλλά παρά τις ε, τόσες συχνές επισημάνσεις, πόρο απέχουμε από αυτήν και αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της ανάπτυξης μιας εσωτερικής αγοράς η οποία θα είναι ανταγωνιστική όπου όπως είπε μόλις και ο συνάδελφος Γιούρ είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ανάπτυξη για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει και αυτή την ενεργειακή αλληλεξάρτηση και τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες ε, για την διαπραγμάτευση με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα λοιπά ε, θα παρουσιάσω μεν κάποιες τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι στο σύνολό της η πρόταση της Εντίτ Herzog είναι πραγματικά καλή και μας επιτρέπει να καθορίσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, τουλάχιστον στα θεμελιώδη ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Τελικαστήγιο. Η κυρία Τόγια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ το λόγο μόνο να, για να προσθέσω μία πτυχή. Η έκθεση της κυρίας Χέρσκο όπως πάντα, είναι πολύ ακριβής και στο προκείμενο. Ε, νομίζω ότι θα παρουσιάσουμε και σχετικές τροπολογίες ε, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης ε, με ταυτόχρονα και τα κατάλληλα νομικά μέσα για να μην είναι υποχρεωτική απαραίτητο, αλλά να είναι πιο ισχυρή συνοχή μεταξύ των κρατών μελών, ιδίω σε μια πτυχή η οποία προβάλλεται εδώ. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένας μόνο ενιαίος αγοραστής όταν αγοράζει ενέργεια από τις ε, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα είχαμε τη δυνατότητα να συνάπτουμε συμβάσεις ε, όχι μόνο από εμπειρική σκοπιάς, αλλά και από ε, σκοπιάς δημιουργίας πιο σημαντικών συμπράξεων και φυσικά η ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν ακόμα πιο ισχυρή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει όλο ένα και περισσότερο ένα ε, ευρωπαϊκό όραμα και όχι ένα διμερές όραμα στις χώρες οι οποίες είναι κυρίως παραγωγή και προμηθευτές ενέργειας και νομίζω ότι αυτό θα ήταν μεγάλο πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θα είναι και η δυνατότητα να εκφράσουμε αυτή την ολοκλήρωση την οποία διεκδικούμε επανειλημμένω στον ενεργειακό τομέα εδώ στην Επιτροπή μας αλλά ε, δυστυχώς υπάρχουν μεμονωμένες δράσεις από χώρες μέλης που είναι ε, εθνικές ε, και ε, μοναχικές εντός εισαγωγικών. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να είναι απλώς κάποιος ο οποίος μιλά με μια φωνή, αλλά θα πρέπει να παρουσιάζεται και με την ισχύ και με μια πιο προφανή στρατηγική δυνατότητα. Με εξέπληξε αυτό που είπε ο κύριος Τούρμες, το ήξερα ήδη, αλλά το να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ λιγότερο στρατηγική στη σχέση της με μια μεγάλη χώρα όπως είναι η Κίνα από ένα κράτος μέλος, σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε στρατηγική όταν υπάρχει βούληση να έχουμε στρατηγική. Εάν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση την επιθυμεί, αυτό θα ήταν σημαντικό για όλε τι χώρε. Την επισημαίνω αυτή την πτυχή γιατί την έχουμε πει επανειλημμένω και επειδή υπάρχουν χώρε προμηθευτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε ε, είναι καταταγμένε και κατά προτεραιότητα, γνωρίζουμε ποιε είναι οι πιο ισχυρέ, θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε μια στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη τη και αυτή την πτυχή. Θεωρώ ότι αυτέ είναι πτυχές οι οποίε θα πρέπει να επισημάνουμε για να ε, δούμε και προς τα πού οδεύει αυτή η εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστώ την κυρία Τόγια. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος να ζητά το λόγο, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυρία Μάρκες. Good afternoon. Thank you very much. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, τις απόψεις που ακούστηκαν εδώ σήμερα. που ενισχύουν ιδιαίτερα την ε, εξωτερική πτυχή της, ε, του ενεργειακού τομέα ε, από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περιμένουμε την τελική εκδοχή του κειμένου. Μας ικανοποιεί ιδιαίτερο το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές υποστηρίζονται τα γενικές ιδέες ε, της ε, πρότασης της ε, Επιτροπής που έγινε το Σεπτέμβριο. Καταρχάς τονίζει το γεγονός ότι η εξωτερική ενεργειακή πολιτική πρέπει να επιτυγχάνει του στόχου της ανταγωνιστικότητας, της αηφορίας και του, της ασφάλειας του ενεργειακού ανεφοδιασμού, όπως επίσης και την εφαρμογή το, του κεκτημένου σχετικά με τον ενεργειακό τομέα. Επίσης, η βελτίωση του συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, σε σχέση με την εξωτερική ενεργειακή πολιτική. Θα θέλαμε να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμό σε σχέση με τις ενεργειακές συμφωνίες με άλλες χώρες, ε, όπως επίσης και μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και επιτροπής για τους τομείς αυτούς. Και αυτό είναι απαραίτητο το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή και να, είναι και πιο, να, παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνοχή οι σχέση της με τρίτες χώρες. Αυτό θα βελτιώσει βέβαια και την ε, ενιαία φωνή που θα έχουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη σε διεθνέ επίπεδο. Μόνο τότε μπορεί να επηρεάσει ε, παγκοσμίω την ενεργειακή ατζέντα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε, έκθεση αναφέρεται όλο ιδιαίτερο στον ενεργειακό ανεφοδιασμό, στην ασφάλειά του και στην ακαιρεότητα τη εσωτερική ενεργειακή αγορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε την εμπειρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην έρευνα, την ανάπτυξη, ε, τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και είναι τομείς ε, προς τους οποίους κινούνται πολλοί εταίροι μας από τρίτες χώρες. Είναι λοιπόν ένας τρόπος να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την συνεργασία και την κατανόηση με τους εταίρους μας οι σχέσεις μας και οι συμφωνίες μας να είναι καλύτερες με τις τρίτες χώρες, είτε είναι αναπτυσσόμενες αυτές είτε είναι ανεπτυγμένες και νομίζω ότι αυτό θα ενισχύσει ιδιαίτερα και θα τονίσει ε, τις, ε, τα θετικά στοιχεία ε, της ε, πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. La parola, la collega... Ευχαριστώ την κυρία Μάρκες. Ε, ο λόγος στην κυρία Μέρκης. Δεν ξέρω αν έχει κάτι να προσθέσει ως αντικαταστάτρια της εισηγήτριας. Τίποτα να προσθέσει, ωραία. Εάν δεν έχετε τίποτα να προσθέσετε λοιπόν... Ολοκληρώθηκε αυτό το τμήμα της συζήτησης. Ε, η συζήτηση επί του περιεχομένου θα συνεχίσει με μια μικρή ακρόαση που θα γίνει αύριο για την ενεργειακή συνεργασία και τις σχέσεις ε, ε, και την εξωτερική διάσταση του ενεργειακού τομέα. Για αύριο το απόγευμα προβλέπεται αυτή η μήνυα κρόση και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχουν συγκεκριμένε προθεσμίες. Ε, κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει ψηφοφορία στην Επιτροπή Ήτρε το Μάρτιο, αλλά ακόμα είναι νωρί για να το οριστικοποιήσουμε. Θα ήθελα τώρα εδώ να κάνω την εξή πρόταση, διότι ήμασταν ε, λίγο πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε προβλέψει. Το τελευταίο σημείο που έχουμε στην ημερήσια διάταξη για σήμερα αφορά το ορίζον 2020 και την κοινή συνεδρίαση με τη δέσμη προτάσεων αυτή και καλό θα ήταν το σημείο αυτό να το ξεκινήσει ο Γενικός Διευθυντής Ρομπέρ Ζαν Σμιθ για να κάνει μια παρουσίαση ε, από την οποία θα ξεκινήσει και η συζήτηση αλλά ο Γενικός Διευθυντής θα είναι εδώ στις 4.30. Προτείνω λοιπόν να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα μισή ώρας, γιατί το να ξεκινήσουμε χωρίς την παρουσίασή τους ε, δεν είναι και πιο λογικό. Είχε προβλεφθεί λοιπόν για τις 4 και μισή. Εμείς τα κάναμε όλα πάρα πολύ γρήγορα, επομένως ε, θα διακόψουμε και θα συνεχίσουμε στις 4 και μισή. Ευχαριστώ πολύ. Ε,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 Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να χαιρετήσουμε λοιπόν τον Γενικό Διευθυντή, τον Ρόμπερτ Ζαν Σμιτ και τον ε, κύριο Κιουρέλ Έχουμε τη χαρά να τους έχουμε εδώ σήμερα για μια συζήτηση για τον ορίζοντα 2020 και ξεκινούμε τις εργασίες μας ε, και να δώσουμε απευθεία το λόγο στο Γενικό Διευθυντή, στο Ρόμπερτ Ζαν Σμιτ, για μια παρουσίαση για τη δέσμη ορίζον 2020. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για την ε, εισαγωγή και καλησπέρα σε όλους. Ε, εδώ με τον συνάδελφο Γιώργη Κουρέλ από την ε, Γενική Διεύθυνση Έρευνας θα σας πούμε λίγα πράγματα για την έρευνα και την τεχνολογία και την κοινοτομία. Παρουσιάστηκε ήδη το Horizon 2020 αμέσως μετά από την ε, έγκρισή του και η Επίτροπος με ενημέρωσε για το πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπήρχε για το θέμα αυτό εδώ στην Επιτροπή σας. Σήμερα θα κάνουμε μια επίσημη ανταλλαγή απόψεων και ελπίζω να είναι η πρώτη μιας μακράς σειράς επαφών και ε, ε, συζητήσεων μεταξύ μας. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την κυρία Σαρτόρη για τον ορισμό της ως πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μαζί σας θα είναι το ίδιο καλή με τον δόκτωρα Ρόιλο, οποίος ήταν ο πρώην πρόεδρος και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την καλή συνεργασία που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ και την κυρία Μαντουρέλ, διότι είναι η συγγήτρια της Επιτροπής ΙΤΡΕ για το Horizon 2020 και βεβαίως θα ήθελα να συγχαρώ και τον δόκτωρα Έλιχ, ο οποίος είναι η συγγητής για τους κανόνες συμμετοχής. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας. Έχω ετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση για το Horizon 2020, το την οποία νομίζω ότι έχετε λάβει όλες. Θα σας πω λίγα πράγματα για το συνολικό πλαίσιο και τη συνολική κατάσταση του Horizon 2020 σε σχέση με άλλες πρωτοβουλίες, το περίγραμμα της πρότασής μας, εγκάρσια ζητήματα και φυσικά το χρονοδιάγραμμα. Καταρχάς, ε, είναι προφανές ότι το Horizon 2020 δεν είναι μεμονωμένο πρόγραμμα, είναι τμήμα του πολιετές δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα παρουσίασε τις προτάσεις της. Πρόκειται για μια πρόταση η οποία καταδεικνύει ότι αφενός ε, χρειάζεται να ε, τακτοποιήσουμε τους διάφορους προϋπολογισμούς, χρειαζόμαστε μέτρα λιτότητας, χρειαζόμαστε δημοσιονομική εξυγίαση, εξυγίανση και ταυτόχρονα χρειαζόμαστε μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν την ανάπτυξη. Πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο μέλλον και όταν αναφερόμαστε σε επενδύσεις στο μέλλον αναφερόμαστε στην παιδεία, στην έρευνα και στην καινοτομία. Για τον λόγο αυτό, αυτό το οποίο μας εντυπωσιάζει, αν δείτε αυτή την πρόταση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει ένας τομέας από όλα τα διαφορετικά πακέτα, τα οποία, ο οποίος λαμβάνει σημαντική αύξηση και είναι ο τομέας της καινοτομίας και της έρευνας. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να υπάρξει μια αύξηση στον προπολογισμό του προγράμματος πλαίσιο ε, κατά 46 περίπου της 100 και αυτό μας οδηγεί σε ένα ε, σύνολο 80 εκατομμυρίων, ε, δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό δείχνει φυσικά πόσο μεγάλη είναι η δέσμευσή μας και πόσο θέλουμε να συνεχίσουμε με μέτρα ε, τα οποία ενισχύουν την ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την Ευρώπη μόνο με μέτρα λιτότητας, πρέπει να υπάρξει και ανάπτυξη και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο προέρχεται από την έρευνα και την καινοτομία. Το Horizon 2020 λοιπόν έχει προχωρήσει, είναι ένα πρόγραμμα ε, συνολικά 80 δισεκατομμυρίων περίπου ευρώ. Όπως σας είπα έχουμε μια αύξηση κατά 46% σε σχέση με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και βεβαίως είναι ένας τρόπος για να ενισχύσουμε τις επενδύσεις στο μέλλον, ώστε να έχουμε μέτρα τα οποία ενισχύουν την ανάπτυξη και να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ανάπτυξη στην οικονομία μας και δημιουργούνται θέσεις εργασίας διασκεδάζει τις ανησυχίες ε, όλων και φυσικά ενισχύει και τη θέση της Ευρώπης παγκοσμίως. Η έκθεση αυτή βέβαια δεν ε, χτίστηκε ε, μέσα από ένα γυάλινο πύργο. Νομίζω ότι αυτή τη φορά πραγματικά ακούσαμε τους ενδιαφερομένους, ακούσαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πραγματικά ε, πριν ετοιμάσουμε την έκθεση αφιερώσαμε αρκετό χρόνο. Έγινε πολύ σημαντική ανταλλαγή απόψεων, για παράδειγμα με την κυρία Καρβάγιο για την απλούστευση, ακούσαμε την κυρία Μερκέση η οποία μας έκανε σημαντικές δηλώσεις για την Ένωση Καινοτομίας και τον κύριο ο ε, Οντί, ο οποίος είχε την έκθεση για την ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του 7ου προγράμματος πλαίσιο και πρότεινε κάτι το οποίο ψηφίστηκε και στην Ολομέλεια, προϋπολογισμό 100 δισεκατομμύριων ευρώ. Δυστυχώ, ε, είμαστε στα 80 δισεκατομμύρια, δεν έχουμε πετύχει ακόμα το στόχο, αλλά φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λόγο, διότι είναι η Δημοσιονομική Αρχή και φυσικά τίναμε και ευήκονου ε, στην έκθεση της κυρία Ματίας ε, για την Πράσινη Βίβλο εν του ορίζον 2020. Τίναμε λοιπόν ευήκονου σε όλες αυτές τις εκθέσεις και φυσικά τίναμε ευήκονου και στους ενδιαφερομένους, το επιστήμονε, στο κλάδο, ε, ακούσαμε και τι προεδρίες, ε, υπήρξε μια ει βάθο ε, διαβούλευση διαδικτυατά, κα, και φυσικά πριν ξεκινήσει λοιπόν η εργασία της εγγραφής της έκθεσης, της εγγραφής της έκθεσης, ακούσαμε όλους ενδιαφερομένους. Εδώ λοιπόν έχουμε κάποιους ε, ένα κατάλογο με τις απόψεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα έχουμε βάλει εδώ στο πίνακα για να δείτε ότι έχουμε συμπεριλάβει τις απόψεις Η, ε, ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής έρευνας και της χρηματοδότησης για την καινοτομία. Εσείς επιμείνατε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η σχέση που υπάρχει με την έρευνα και την ε, ε, καινοτομία και είπατε ότι πρέπει να τη συνδέσουμε και το κάναμε. Ζητήσατε μια εκβάθρον απλούστευση. Η κυρία Καρβάγιο πίεσε προς αυτή την κατεύθυνση και εμείς προτείνουμε μια εκβάθρον απλούστευση και εδώ η κυρία Καρβάγιο μας λέει ότι ίσως υπεραπλουστεύσαμε τα πράγματα αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό εντός ολίγου. Ε, βασική επιστήμη. Πολύ σαφές δηλώσεις και από, και από τον κύριο Ρόιλ αλλά και από άλλους στο παρελθόν πρέπει να, αρχίσουν, να αρχίσουμε να επενδύουμε σε βασική έρευνα και βλέπετε ότι έχουμε ένα εντυπωσιακό ε, πακέτο για να ενισχύσουμε αυτή τη βασική επιστήμη, τη βασική έρευνα ιδίως στον τομέα του ERC που ήταν πολύ σημαντικό και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επικεντρωθούμε στις προκλήσεις της κοινωνίας. Εάν υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο προέκυψε σαφώς από την έκθεση της κυρίας Ματίας είναι να διασφαλίσουμε ότι θα ε, επικεντρωθούμε στις ε, προκλήσεις της κοινωνίας, θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες των πολιτών και φυσικά οι ανησυχίες των πολιτών αφορούν την υγεία τους, την ασφάλειά τους, τα τρόφιμα που καταναλώνουν, τις μεταφορές και ούτω καθεξής. Επομένως, Έχουμε περάσει από μια θεματική προσέγγιση ε, που μας πίεζε η τεχνολογία να καταλήξουμε στο να εισακούσουμε τι έχουν να μας πούνε οι πολίτες. Επίσης, ε, ε, πολλαπλή συμμόρφωση, πολλαπλές επιστήμες και αυτό το έχουμε στην πρότασή μας. Σε αρκετές περιπτώσεις έγινε συζήτηση εδώ για το κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε ευρύτερη συμμετοχή ο κύριος Έιλερ και η κυρία Τζόρντεν ασχολήθηκαν με τα θέματα αυτά και ε, διασαφήνισαν ότι είμαστε μια Ευρώπη των 27 και ότι η αριστεία υπάρχει παντού και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ε, η αριστεία ακόμα και σε χώρες οι οποίες δεν εκπροσωπούνται και τόσο καλά στο ε, πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν. Επομένως ε, κάνουμε κάποια ενδιαφέροντα ε, μέτρα για να διευρύνουμε τη συμμετοχή ε, χώρεων και οργανώσεων στο πρόγραμμα πλαίσιο. Επιπλέον, και αυτό το είχαμε και στην έκθεση της κυρίας Ματίας, υπάρχει το γεγονός ότι η καινοτομία δεν είναι μόνο τεχνολογική καινοτομία, αλλά και κοινωνική καινοτομία. Ακούσαμε λοιπόν τι έχετε να μας πείτε και θα δείτε ότι στην πρότασή μας στο Horizon 2020 ασχολούμαστε με το θέμα της ε, κοινωνικής καινοτομίας. Και επίσης ε, ε, κάτι εξίσου σημαντικό, το οποίο ζητήσατε πολλοί από εσά, ε, τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τον κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και εμείς στο ορίζον 2020 κάνουμε μια εντυπωσιακή πρόταση και με χρηματοοικονομικά μέτρα και με προπολογισμό για να υπάρξει στήριξη στις επιχειρήσει. επιχειρήσεις. Δεν είναι εδώ ο υπεύθυνο, διότι είναι ε, στην Επιτροπή Προπολογισμών και συζητάει τα θέματα τη απαλλαγή. Το Horizon 2020 βασίστηκε σε τρεις βασικές προτεραιότητες. Άριστη επιστήμη, ε, βιομηχανική ηγετική θέση και ο ρόλος της κοινωνίας. Γιατί θέλουμε να έχουμε άριστη επιστήμη. Αυτό νομίζω ότι είναι προφανές. Εάν δεν επενδύσουμε ευθύ εξ αρχής ε, ε, στην ε, επιστήμη δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την επιστημονική της βάση. Θα πρέπει να επενδύει σε μεγάλες κλίμακες εγκαταστάσεις όπου μπορούμε να ελοπίσουμε το έργο μας και επιπλέον θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να ενισχυθούν, να τους επιτρέψουμε να κάνουν βασική έρευνα και να έχουν και κινητικότητα και να μετακινούνται στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό ακριβώς ε, δίνουμε προτεραιότητα στην ενίσχυση της άριστης επιστήμης διπλασιάζεται σχεδόν ο προπολογισμό ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνα. Το ERC ήταν μία από τι επιτυχημένε ιστορίε του προγράμματο πλαίσιο και αναγνωρίστηκε και από την Επιτροπή σα, ε, υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εγγέννη. Σα ανέφερα ήδη την κυρία Νίπλερ, θα έπρεπε να αναφέρω και την κυρία Γκροστέτ, αλλά και πολλού άλλου οι οποίοι υποστηρίζουν αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία και προτείνουμε να διπλασιαστεί σχεδόν ο προπολογισμό τη ε, μελλοντικέ και αναδυόμενε τεχνολογίες. Κυρία Καρβάγιο, πριν από δύο χρόνια ζητήσατε να εισηχθεί αυτό και να ενισχυθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα και αυτό γίνεται και μάλιστα με ουσιαστικό τρόπο Δράσεις Marie Curie, πάρα πολύ σε ένα πρόγραμμα κινητικότητα, πολύ δημοφιλέ μεταξύ των νέων ερευνητών και σίγουρα θα ενισχυθεί και αυτό. Και τέλο, εξίσου σημαντικέ, ε, οι βασικέ υποδομές. Όπω σα είπα, είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη να προετοιμαστεί για την επόμενη γενεά ε, υποδομών, δηλαδή ε, υποδομέ μεγάλη κλίμακα, οι οποίε να είναι ανοιχτέ σε ερευνητέ από όλη την Ευρώπη, ώστε πράγματι να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε προωθήσουμε τη γνώση της επιστήμης. Υπάρχει λοιπόν εντυπωσιακό προπολογισμό για αυτό τον πυλώνα τη αριστεία. Επίση, θα πρέπει να ενισχύσουμε τον ηγετικό μα ρόλο στη βιομηχανία. Στην έκθεση του κυρίου Οντί για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του 7ου προγράμματο πλαίσιο, ε, φάνηκε πολύ σημαντικό ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Και εδώ ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, μέσω αυτού του πυλώνα της ηγετικής θέσης στη βιομηχανία, γιατί θέλουμε η βιομηχανία να επανέλθει στα προγράμματά μας. Είδαμε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια ότι έχει μειωθεί η συμμετοχή του βιομηχανικού κλάδου και νομίζω ότι ήγηκε η ώρα να επανέλθει και πάλι στα προγράμματα πλαίσιο, διότι δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της έρευνας και της καινοτομίας και τα όσα προβλέπει και η συνθήκη της Λισαβόνας είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο προς αυτό το πλαίσιο και θα δείτε ότι πέραν από τις επενδύσεις και τις τεχνολογίες που είναι βασικές, έχουμε 13 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις, έχουμε και ένα σημαντικό πακέτο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 15% του προπολογισμού για τις προκλήσεις για την κοινωνία θα το αφιερώσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θέλουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία του Eurostar, η οποία ε, συμβαδίζει με το Eureka και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και συνέχεια ε, του Risk Finance Facility. Ε, υπήρχαν αρκετές δραστηριότητες προς αυτό το τονέο και με χαρά θα διαπιστώσετε ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση κινδύνου θα συνεχιστεί στο Horizon 2020. Ο τομέας της ε, χρηματοδότησης ε, κινδύνου είναι και πάλι ένα επιτυχημένο ε, τμήμα. Είχαμε και μία παρουσίαση της Έρικα Μαν για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση αυτής της δυνατότητας και η έκθεση αναγνώριζε ότι και ήταν επιτυχημένη και επίσης με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι ακόμα και μόλις μετά από δύο χρόνια λειτουργία αυτού του μέσου σχεδόν 8 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν ω επιδότηση σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Επομένως, εκτός από ανάπτυξη υπάρχει και αγορά για επιδότηση σε επιτυχημένα προγράμματα. Ήδη ανέφερα ότι ε, διαπιστώσαμε ε, ότι χρειάζεται να αναφερόμαστε στο μέλλον στις ανάγκες της κοινωνίας και όντως εδώ σκεφτήκαμε μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση και προσπαθούμε έτσι να διασκεδάσουμε τις ανησυχίες των πολιτών. Και εδώ αναφέρομαι στην ε, ανησυχία για την υγεία, για την, ε, τα τρόφιμα, για το κλίμα και βεβαίως ο, ο πολίτης θέλει να ζει σε μια ασφαλή κοινωνία. Είναι προφανές ότι αυτές οι προκλήσεις είναι προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, και μέσω των των βιομηχανιών και μέσω των ε, ερευνητικών εταιριών θα χρειαστεί συνεργασία για να μπορέσουν να δοθούν λύσεις που θα ικανοποιούν τους πολίτες. Και αυτό χρειάζεται διότι στον τομέα της υγείας είδαμε ότι η μελέτη απέδειξε ότι σε λίγο η ε, γεροντική άνοια θα ε, κοστίζει τεράστια ποσά για την Ευρώπη και πέραν της ανθρώπινης τραγωδίας που αντιπροσωπεύει. Πρέπει λοιπόν στην Ευρώπη να ενώσουμε τις δυνάμεις ε, μας και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη φοβερή ασθένεια, το Αλτσχάιμερ και την Άνια και να μπορέσουμε να προσφέρουμε λύσεις. Πέραν αυτού, όσον αφορά τις κοινωνικές επιστήμες, ε, παίζουν ένα βασικό ρόλο ε, τις τις ε, προκλήσεις ε, που τίθενται στην κοινωνία και αποτελούν μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με την ισχύουσα κατάσταση. Δεν σκοπεύουμε με διαφορετικό πρόγραμμα για τις κοινωνικές επιστήμες ε, και ε, τη γενική μόρφωση, αλλά εφόσον ε, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την φυσική και για τη χημεία, γιατί να έχουμε για τις πολιτιστικές επιστήμες. Η πρότασή μας λοιπόν είναι η εξής, ότι οι κοινωνικές επιστήμες μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην επίλυση των προκλήσεων της κοινωνίας αρκεί ε, να εξετάσουν και να επεξεργαστούν τα βασικά προβλήματα της κοινωνίας στον τομέα της υγείας. Διάβασα ορισμένες στατιστικές για τη χώρα μου την Ολλανδία το περασμένο Σαββατοκύριακο όπου έλεγε ε, ότι ε, ένα ακόμα οκτώ άτομα έχει μόνο μία επαφή το μήνα στη μεγάλη ηλικία στην οποία βρίσκεται. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα για τις κοινωνικές επιστήμες. Πρέπει να επιλύσουν την απομόνωση αυτή. Εάν λοιπόν αλλάξουμε το πρόγραμμα, χωρίς να αλλάξουμε λοιπόν το πρόγραμμα, τους λέμε σας προκαλούμε καλούμε να αλλάξετε τη δομή της κοινωνίας, να αναλάβετε τις ευθύνες σας, να συμβάλλετε στην εξέβρεση λύσεων για όλες τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Είναι κάτι προκλητικό, αλλά μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ε, ε, είναι πολλές βέβαια δραστηριότητες, αλλά με το ε, ERC, το Ευρωπαϊκό δηλαδή Συμβούλιο Ερεύνης, μπορέσαμε να διαθέσουμε 70% των πόρων για την έρευνα στον κοινωνικό τομέα, άρα αυτό είναι πολύ θετικό. Σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ήδη ανέφερα ότι αποβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτές θα συμπεριληφθούν στα προγράμματα όταν θα έχουν απλοποιηθεί και θα υπάρχει ένα πρόσύστημα που θα έχουμε αντιγράψει από τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, χρησιμοποιώντας το πρότυπο SBIR πράγμα το οποίο θα τους επιτρέψει να έχουν μελέτες σκοπιμότητος δωρεάν και τέλος θα μπορέσουμε ε, να, τους, να τις στηρίξουμε μέχρι να προωθηθούν τα ε, προϊόντα τους στην αγορά. Πράγμα το οποίο γίνεται στι Ηνωμένε Πολιτείε και σε διάφορα κράτη-μέλη και έφτασε η ώρα κάτι τέτοιο να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε επίσης να υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο θα χρηματοδοτούμε και το ενεργητικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, να υπάρχει μια διευρυμένη συμμετοχή διότι όπως ανέφερα είμαστε μια Ευρώπη των 27 και σύντομα 28 κρατών μελών. Πρέπει λοιπόν όλες οι ερευνητικές ομάδες των κρατών μελών που είναι εξαιρετικές να ενταχθούν στα προγράμματά τους γιατί πολλές φορές η αριστεία κρύβεται και πρέπει να την προβάλλουμε και να, την, να ε, της δώσουμε τη θέση που χρειάζεται στα προγράμματά μας. Γι' αυτό και αποδίδουμε μεγάλη μεγάλη σημασία στη δυνατότητα των χωρών να μπορούν να αναπτύξουν τις δυνατότητες αριστείας και προωθήσεως προγραμμάτων και αυτό μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Ο κύριος Βανίσελ Ρόι συνεργάστηκε ε, και στο παρελθόν για τα προγράμματα πλαίσιο και ε, προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε εφαρμόσουμε τα προγράμματα αυτά με τον εξή τρόπο. Τα διαρθρωτικά ταμεία θα χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν την έρευνα και την τεχνολογία, να μπορούν οι χώρες να εξυγχρονίσουν τα πανεπιστήμια, να προσλάβουν προσωπικό και ο ρόλος του ορίζοντα 2020 είναι να τονίσει την ευρωπαϊκή αριστεία και η συνεργασία αυτή θα ενταθεί διότι πρόκειται για δύο βασικά μέσα χρηματοδότησης για να μπορούμε όπως σας είπα να προωθήσουμε την αριστεία και να προωθήσουμε ε, ε, τις εξαιρετικές ε, προσωπικότητες μέσω του προγράμματος Ορίζοντες 2020. Έτσι το, στηρίζουμε την αριστεία η οποία δεν θα περιοριστεί μόνο σε ορισμένα σημεία της Ευρώπης αλλά θα επεκταθεί και περαιτέρω. Διεθνή συνεργασία. Πολλά μέλη αυτής της Επιτροπής μας έχουν τονίσει επανειλημμένως ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι απομονωμένη αλλά να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής σε προσπαθίας να μην έχουμε ένα οχυρό Ευρώπης. Οπότε στον ορίζοντα 2020 προσπαθήσαμε να διευρυνθούμε στη συμμετοχή όλων των χωρών του κόσμου. Ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ορίζον 2020 βάσει αριστείας και βάσει της δεδηλωμένης επιθυμίας της Ευρωπαϊκής ε, ε, ε, ενώσεως να συνεργαστεί με τις τρίτες χώρες, δηλαδή ε, θα προωθήσει την συνεργασία όπου χρειάζεται με την Νότιο Αφρική, με την Νότιο Κορία, με την Ασία, διότι μόνο έτσι θα προχωρήσουμε. Και πάλι θα συνεχίσουμε με τις συμφωνίες συνδέσεων. Έχουμε πολλές χώρες όπως η Ελβετία και η Νορβηγία που συνδέονται και το ορίζο 2000 2020 θα επιτρέπει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με συνδεδεμένες χώρες. Δεν θα αναφερθώ ή στον ρόλο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ε, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, EIT, γιατί αυτό θα το ε, παρουσιάσει ο διπλανός μου, αλλά προσπαθούμε να έχουμε μία σωστή ε, επιστημονική βάση και για αυτό το κοινό ε, ερευνητικό κέντρο είναι η βάση του προγράμματος Horizon 2020. Κυρία Καρβάλιο, διαβάσαμε επανειλημμένο στην έκθεσή σας για να εξασφαλίσουμε ότι θα απλοποιήσουμε το τέρας αυτό που ήταν το καρκίνωμα του προγράμματός μας. Τώρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει ριζική ε, απλοποίηση και θα έχουμε απλούς κανόνες. Μόνο ένα σύνολο κανόνων που θα είναι ε, ένα πρόγραμμα με ένα ποσοστό συμμετοχής θα έχουμε απλούστερες μεθόδους χρηματοδοτήσεως και ε, νέες μορφές συνεργασίες, πιο απλούς κανόνες ε, για τις χορηγήσεις, λιγότερους ελέγχους ελέγχους και ε, βελτιωμένους κανόνες για την πνευματική ιδιοκτησία κατά τρόπον ώστε οι προσπάθειές μας να απλοποιήσουν ριζικά το σύστημα. Πήρα τον ε, κατάλογό σας κυρία Καρβάλιο και έχω σημειώσει τι κάναμε. Βλέπετε λοιπόν ότι σε όλα τα σημεία ακολουθήσαμε τις συστάσεις σας. Εσείς μπορείτε να μας πείτε ε, που κάτι μας ξέφυγε ή που το παρακάναμε γιατί ξέρω ότι εσείς όπως και η κυρία Φόρντ αναφέρθηκαν στο οικονομικό κόστος των τροφίμων αλλά θα επανέλθουμε μαζί με τις παρατηρήσεις του κύριο Βαλνίστερ Ρόι στα θέματα αυτά. Θέλω το Κοινοβούλιο να μας στηρίξει σε αυτή την κατεύθυνση διότι οι ε, κανόνες ήταν πολύ περίπλοκοι, μας διακατήχει η προσπάθεια των τελείων ελέγχων αλλά δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, δηλαδή σωστή έρευνα και δεν πρέπει ο έλεγχος να παρεμβαίνει στην ερευνητική εργασία. Βέβαια να υπάρχει σωστή δημοσιονομική παρακολούθηση και θέλουμε <clears throat> να μπορέσουμε να βρούμε μία σωστή ισορροπία μεταξύ των διαφόρων παραμέτρων για την, μεταξύ της έρευνας και της οικονομικής διαχείρισης. Πώς όμως θα συνδυάσουμε ε, το ε, ορίζοντα 2020 με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ερεύνης. Ε, θα κοιτάξουμε την δυνατότητα μεταφοράς των χορηγήσεων, κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί από τα εθνικά ερευνητικά συμβούλια. Θα πρέπει να ε, υπάρξει ε, διαφάνεια στα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Μπορούν εκεί να μας στηρίξουν και τα κράτη-μέλη αλλά και οι εθνικές οργανώσεις που θα στηρίξουν το ERA και μιλάμε για το πρόγραμμα κινητικότητος, μιλάμε ε, και για άλλες δυνατότητες και αναλαμβάνουμε τις ευθύνες Έλληνες μας κατά τρόπον ώστε ο ορίζον 2020 να δημιουργήσει εξελίξεις στο χώρο της έρευνας. Έχουμε και μία πρόταση για την Ευρατόμ. Ε, την ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ε, κυρία Χέρσο από αυτό, ε, ειδικότερα ό,τι έχει να κάνει με την Ευρατόμ. Πρόκειται να τονίσουμε ιδιαίτερα την πυρηνική ασφάλεια και την κατάρτιση για τα πυρηνικά θέματα για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε αρκετή τεχνογνωσία για τον παροπλισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων και ότι έχουμε αρκετούς ε, ειδικού ε, για την προστασία από την ακτινοβολία και για την ε, πυρηνική ασφάλεια. Αν, και ειδικότερα αν θέλουμε να καταργήσουμε σταδιακά τους πυρηνικούς αντιδραστήρες μας. Εκτός από το πρόγραμμα Horizon 2020 έχουμε και το πρόγραμμα COSME ε, υπάρχει βέβαια μια μεγάλη, μια έντονη σύνδεση μεταξύ ε, του δικού μας προγράμματος του Ορίζοντα 2020 και του κόσμου για να εξασφαλίσουμε με τους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση ε, ε Βιομηχανίας ότι υπάρχει πλήρη συμπληρωματικότητα των ε, δύο δράσεων. Φτάνω σιγά σιγά στο τέλος της παρουσίασής μου, συγγνώμη που μακρηγόρησα τόσο. Θα γίνει μια βάθο συζήτηση μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζουμε ότι περίπου κατά τα μέσα του 2013 θα καταλήξουμε έτσι σε έγκριση των νομοθετικών πράξεων που δίνουν την ε, έγκριση ε, στον ορίζοντα 2020 ε, ώστε να αρχίσουμε τις, τους πρώτους μας διαγωνισμούς τον Ιανουάριο του 2014. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και για όλα τα σχόλιά σας ε, ελπίζω να σας έδειξα και στην παρουσίασή μου ότι σας ακούσαμε πραγματικά και εξακολουθούμε να θέλουμε να σας ακούμε σε σημεία που δεν σας βρίσκουν σύμφωνους ή θεωρείτε ότι δεν ελήφθησαν υπόψη επαρκώς τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον Ρόμπερτ Τζαν Σμιθ και τώρα να δώσουμε το λόγο στον ε, Διευθυντή Ζορντί Κουρέλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια και από δική μου πλευράς για τον ε, ε, διορισμό σας. Θα ήθελα να συγχαρώ και τους δύο εισηγητές, ε, τις δύο εισηγήτριες για τι πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία προκειμένου να είναι καρποφόρα η προσπάθειά μας αυτή. Τα καλά νέα ε, είναι ότι επιτέλους το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, το EIT, ε, έχει βρει τη θέση του, δεν είναι πλέον το ορφανό ε, στην, στο, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έχει βρει λοιπόν μια θέση είναι ένα τμήμα του ορίζοντα 2020, του προγράμματος αυτού. Και θα ήθελα να μην σας διαφεύγει αυτό, γιατί η, βασική, η βασική κατεύθυνση που είχαμε εμείς ε, ε, όταν υποβάλαμε την πρόταση αυτή ήταν ακριβώς να εξασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας θα συνέβαλε στους στόχους του ε, ορίζοντα 2020 αλλά και της στρατηγικής για το 2020. Οι διατάξεις λοιπόν για την παρακολούθηση, ε, για την αξιολόγηση θα ισχύουν και για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και για το θέμα της απλοποίησης. Ε, οι κανόνες του ορίζοντα 2020 θα ισχύουν και για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ε, με τις απαραίτητες βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν βέβαια σε σχέση με την εφαρμογή των κανόνων αυτών. Για ποιο λόγο βρισκόμαστε όμως εδώ σήμερα. Είμαστε εδώ σήμερα με την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί η αρχική ιδέα που ήταν ε, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία, ο λόγο ύπαρξή του, εν πάση περιπτώσει, βρήκε επιτέλου. Ε, ε, παίρνει επιτέλου σάρκα και οστά. Έχουμε λάβει υπόψη σημαντικές συνεισφορές, για παράδειγμα, ε, το, την agenda που προτείνει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο και ε, τη λάβαμε βέβαια το Μάιο του 2011, την εξετάσαμε πολύ προσεκτικά και θα δείτε ότι υπάρχει μεγάλη σύγκληση μεταξύ του τι προτείνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο και το τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ινστιτούτο. Ε, Υπήρξε επίση και μια ανεξάρτητη αξιολόγηση, είναι στη διάθεσή σας αν, ε, την, ε, αν επιθυμείτε να τη διαβάσετε. Και πήραμε και κάποια μαθήματα από την αξιολόγηση αυτή. Υπάρχουν πολύ σημαντικά σημεία, υπάρχουν, πολύ, υπάρχουν σοβαρά, ε, σοβαρές, σοβαρά ισχυρά σημεία ε, στον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Γενοτομίας και Τεχνολογίας, αλλά υπάρχουν δυστυχώς και κάποιες αδυναμίες. Έγινε και μία συζήτηση με εμπλεκόμενους φορείς, ε, υπήρξαν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ε, τις εξετάσαμε και αυτές ε, όλος ιδιαιτέρως. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να αρχίσω με τις προτεραιότητες του Ινστιτούτου. Όπως είπα και προηγουμένως, η βασική προτεραιότητα είναι η συνεισφορά στους στόχους ε, του ορίζοντα 2020 μέσω των κοινοτήτων ε, ε, καινοτομίας και γνώσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που προτείνουμε είναι το Ινστιτούτο να παγιώσει ε, τις υπάρχουσες πληροφορίες μέσω ανταγωνιστικών μηχανισμών ώστε να υπάρχουν ε, να υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης ε, από τους ε, ομοτήμους προκειμένου να βελτιωθεί η ολόκληρη, η διαδικασία. Επίσης προτείνουμε τα εξής. Προτείνουμε καταρχάς να, υπάρχει, να υπάρχουν τρία νέα προγράμματα το 2016 και άλλα τρία το 2018. Θα επανέλθουμε ούτω ή άλλω με περισσότερε λεπτομέρειε όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τον προπολογισμό και του μηχανισμού αναθεώρηση ε, για το δεύτερο τμήμα ε, δρομολόγηση προγραμμάτων. Αυτό που προτείνουμε, όπως θα είδατε άλλωστε, είναι ότι ε, υπάρχει επικάλυψη με, τα με τις θεματικές ενότητες του ορίζοντα 2020 και αυτό είναι λογικό γιατί είμαστε τμήμα της μεγάλης αυτής οικογένειας πλέον και πρέπει να συνεισφέρουμε στην επίτευξη των στόχων της. Τα τρία ε, τωρινά προγράμματα που αφορούν ε, την αηφόρο ενέργεια από τη μία, την κλιματική μεταβολή και ε, την τεχνολογία της ε, πληροφορίας. Προσπαθούμε ε, να έχουμε και ένα πρόγραμμα για την καλύτερη διαβίωση, για, τα, για τις πρώτες ύλες και το 2018 προστιθέμενη αξία για την μεταποίηση και την αστική κινητικότητα. Όσον αφορά λοιπόν τη θεματική ε, ενότητα των κοινωνικών προκλήσεων ε, είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε γιατί υπάρχουν διάφορες οπτικές γωνίες από τις οποίες μπορεί να ειδωθεί το θέμα και προσπαθήσαμε να γίνει μια διεξοδική ανάλυση στην δική μας ε, στρατηγική ατζέντα καινοτομίας δείχνουμε ότι έχουμε λάβει υπόψη το κατά πόσο μια θεματική ενότητα ε, πρέπει να ε, αντιμετωπίζεται ως τέτοια ή όχι. Και στη συνέχεια αυτό το υποβάλαμε σε ε, διαβούλευση. Είναι πάρα πολύ εμφανές αυτό στην πρότασή μας και γι' αυτό ακριβώς το συγκεκριμένο κείμενο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό προϊόν. Βέβαια, θα συζητηθεί, πρέπει να συζητηθεί, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ σοβαρής ε, και λεπτομερούς δουλειάς και ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι καλό είναι να το συζητήσουμε με λεπτομέρεια. Και το λέω αυτό γιατί στον τρέχοντα κανονισμό, όπως γνωρίζετε όλοι, οι θεματικές ε, ενότητε, ε, η κλιματική μεταβολή, η αιφορό ενέργεια και ε, η τεχνολογία της πληροφορίας, νομίζω ότι είναι ζητήματα τα οποία ε, είναι ε, ενδιαφέροντα για όλους και γι' αυτό πιστεύω ότι η διαδικασία ήταν ικανοποιητική. και γι' αυτό πιστεύω ότι και ο στόχος μας ε, θα επιτευχθεί με ικανοποιητικό τρόπο. Η δεύτερη προτεραιότητά μας ε, θα είναι κάτι πέρα από τα προγράμματα αυτά, δηλαδή πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας πρέπει να εστιάσει τους ανθρώπους, πρέπει να ενισχύσει τον αντίκτυπό του εστιάζοντας στους ανθρώπους και αναζητώντας ταλαντούχους ανθρώπους. Επομένως θα υπάρξει ένα πρόγραμμα fellowship του, ε, με σκοπό να διευκολυνθεί η ανταλλαγή ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων ε, ε, και βέβαια θα, ε, θα οικοδομηθεί έτσι και μία κοινότητα πρώην μαθητευομένων στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο. Πρέπει να δούμε λοιπόν ότι Πρέπει να δούμε και την ευελιξία των κανόνων. Δηλαδή, πρέπει να προβλέψουμε για το Ινστιτούτο τη δυνατότητα να μην είναι γραμμένα τα πράγματα στην πέτρα μέχρι το 2020, αλλά να υπάρχει κάποιο είδου ευελιξία ώστε να μπορέσει να ε, αντιμετωπίσει προβλήματα και προκλήσεις που θα προκύψουν. Τώρα, Πώ πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Πρώτον, είναι ένα ζήτημα προπολογισμού. Χρειαζόμαστε χρήματα για να κάνουμε οτιδήποτε. Βλέπετε ότι η Κομισιόν έχει προβλέψει έναν προπολογισμό περίπου 3,2 δισεκατομμύρια για ολόκληρη την περίοδο. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί και στο Κοινοβούλιο σε μεγάλο βαθμό, ε, γιατί εσεί έχετε σχεδόν τον τελευταίο λόγο από κοινού με το Συμβούλιο και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πρέπει όμως να ε, συζητήσουμε πέρα από το ποσό που προτείνεται αυτή τη στιγμή. Είπαμε ότι είναι τμήμα του ευρύτερου πακέτου των 80 δισεκατομμυρίων και πρέπει νομίζω να συζητήσουμε τον ε, ειδικό μηχανισμό που έχουμε εφεύρει προκειμένου να ε, αποδεσμεύονται αυτά τα κονδύλια. 3,2 δισεκατομμύρια για όλη την περίοδο. Ελπίζουμε να είναι δύο τα κομμάτια, 2,5 δισεκατομμύρια στην αρχή ε, μέχρι το 2014 και από το 2014 μέχρι το 2017 για τα ε, προγράμματα και για τα τρία νέα προγράμματα που θα αρχίσουν το 2014. Με το τέλος του 2017 η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση και θα, θα εξετάσουμε ακριβώς αυτό, κατά πόσο χρησιμοποιήθηκε σωστά ε, ο προϋπολογισμός και είχε και αρκετό αντίκτυπο από τη μία πλευρά και επίσης πρέπει να εξετάσουμε και τα ε, χρήματα που θα ε, αποδεσμευθούν μετά για τα υπόλοιπα προγράμματα. Αν θεωρήσουμε ότι όντως ε, πληρούνται οι προϋποθέσεις, ε, τότε θα εκταμιευθεί το επόμενο ποσό του 1,6 δισεκατομμυρίου για το, την περίοδο 2017 έως 2020. Το τελικό σημείο που θα ήθελα να δείξω και νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρώσω εδώ γιατί το σημαντικότερο τμήμα είναι η ερωταποκρίση σε τέτοιου είδους συζητήσεις, είναι να συζητήσουμε λοιπόν λοιπόν ε, να δούμε το θέμα της εμπειρίας, ε, της αξιολόγησης, ε, της ανεξάρτητης αξιολόγησης που έγινε και καταλήξαμε σε κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης του Ινστιτούτου. Δεν θα πω σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί πιστεύουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα έπρεπε να είναι λίγο μικρότερο ε, να αριθμεί λιγότερα μέλη για να είναι πιο ευέλικτο. Και γι' αυτό προτείνουμε ένα φόρουμ ε, stakeholders του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για να εξεταστούν ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Η τελευταία πρωτοβουλία στον τομέα αυτό είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν ακόμη περισσότερες συνέργειες μεταξύ του Ινστιτούτου ε, των προγραμμάτων και οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας ε, την οποία έχουμε εξετάσει. Καλό είναι να σταματήσω εδώ νομίζω. Ελπίζω αυτό να σας έδωσε μια γενική εικόνα της πρότασης που έχετε ε, νοποιών σας και αν έχετε τυχόν ερωτήσεις ευχαριστώ να απαντήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. συμφωνήσαμε με τους δύο γενικούς διευθυντές να γίνει ένας πρώτος γύρος ε, παρεμβάσεων με τους εισηγητές και κατόπιν θα ήθελαν να δώσουν μια πρώτη απάντηση, μετά να ακούσουμε τους κοιόδης εισηγητές ε, μια δεύτερη απάντηση και από εκεί και πέρα έχουν όλοι το λόγο ελεύθερα, διότι θεωρούν ότι το θέμα ε, πρέπει να χωριστεί έτσι, θα ήταν πιο χρήσιμο. Ξεκινούμε λοιπόν με του συζητητέ. Από πέντε λεπτά ο καθένα. έχουν ζητήσει πάρα πολλοί συνάδελφοι το λόγο. Πραγματικό λοιπόν θα θέλαμε να σα ζητήσουμε να σεβαστείτε τα χρονικά περιθώρια. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Μαντουρέλ. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σμιτ και ευχαριστώ και τον κύριο Κουρέλ διότι ήρθατε εδώ για να μας παρουσιάσετε αυτό το σημαντικό πακέτο προτάσεων, αυτή τη δέσμη ε, και το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για τον ορίζοντα 2020. Σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια για μένα. Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε πολύ στενά, ιδίως ε, για τα θέματα αυτά στους επόμενους μήνες. Επομένως, ε, όπως λέει και ο Χάμφρι Μπόγκαρτ, πιστεύω ότι αυτή είναι η αρχή μιας υπέροχης φιλίας. Νομίζω ότι ε, πρέπει να καθορίσουμε και τις θέσεις μας, μας περιμένει πολλή δουλειά, αλλά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι συμφωνούμε με την ανάλυση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις περισσότερες από τις αρχές ε, που βρίσκονται στη βάση αυτού του τόσο σημαντικού ζητήματος. Για παράδειγμα, συμφωνούμε ότι είναι πολύ περίπλοκο το σύστημα έρευνας και καινοτομία, αλλά για να μεταφράσουμε από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα σε προϊόντα είναι πολύ μεγάλες δυσκολίες και από εκεί και πέρα θα πρέπει να αποτελέσουν όλα αυτά στόχο για την ανάπτυξη όπως εξηγήσατε και εσείς και αυτό επίσης συμφωνούμε. Να σας πω απλώς ότι η ομάδα μου υποστηρίζει την ιδέα του ορίζοντα του 2020 ως το πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει όλη την αλυσίδα της καινοτομίας από τη βασική έρευνα ε, μέχρι την αγορά και την επικέντρωσή του σε μια e e, ευφυή ανάπτυξη που θα συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Και επειδή ακριβώς αυτό το πρόγραμμα ανάπτυξης ε, γεννάται στη συγκυρία αυτής της ε, κρίσης με πολύ σοβαρούς περιορισμούς των προπολογισμό στα περισσότερα κράτη-μέλη, υπάρχουν ε, κάποια στοιχεία τα οποία μα ανησυχούν και θα ήθελα να θέσω ευθύ εξ αρχή. Το πρώτο ζήτημα που μα ανησυχεί είναι πώ μπορούμε να αποφύγουμε στο μέλλον να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη πόλωση του επιστημονικού και τεχνολογικού μας χάρτη ε, του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού και Τεχνολογικού Χάρτη. Πρόκειται για κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρο αν θέλουμε να προχωρήσουμε ορθώς ε, στην ε, δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Συμφωνούμε όλοι ότι ιδίω όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα για, το μεγαλύτερο συντονισμό και ούτω καθεξής θα πρέπει να δώσουμε τη δέωση σημασία στα μέσα τα οποία επιτρέπουν τη συμμετοχή ε, στο χάρτη των διαφόρων κρατών μελών. Δηλαδή ε, συμμετοχή ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, τις δυνατότητές τους και τις συνάφειές τους. Θεωρούμε όμως ότι αυτή τη στιγμή μια τέτοια τοποθέτηση μπορεί να μην είναι απόλυτα ρεαλιστική διότι μπορεί να μας οδηγήσει όπως σας είπα ε, προηγουμένως, σε μεγαλύτερη πόλωση του επιστημονικού και τεχνολογικού χάρτη της Ευρώπης. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να αποφύγουμε τη μεγαλύτερη πόλωση χωρίς να ξεκινήσει η συζήτηση της ε, εδαφικότητας ενός προγράμματος και να μην απαρνηθούμε φυσικά και την αριστεία που είναι ο στόχος μας. Εσείς επίσης λέτε ότι οι πολιτικές συνοχές θα πρέπει να προσφέρουν ε, μια κλίμακα προς την αριστεία και για μένα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ε, μια πολύ ωραία εικόνα την οποία θα πρέπει να εμβαθύνουμε και θα ήθελα να ξέρω κάποια περισσότερα στοιχεία για το πώς ε, βλέπει αυτή την κλίμακα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πραγματικότητα. Τι ακριβώς έχετε κατά νου, πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να οικοδομηθεί, από ποια υλικά. Ε, τι ε, είδους ε, υλικά θα χρησιμοποιήσουμε, τι προτεσίλες. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό, διότι το βασικό ζήτημα είναι πώς θα έχουμε συνέργειες με τα άλλα προγράμματα. Πρόκειται για κάτι το οποίο συζητήθηκε ιδιαίτερα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και πρόκειται για μια συζήτηση η οποία είναι ακόμα πιο σημαντική αυτή τη στιγμή διότι βιώνουμε κρίση και ε, θα πρέπει να αναγνωρίσω εδώ ότι ο ορίζοντας 2020 αποτελεί μεγάλη πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Καταφέραμε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή συνέργεια με το πρόγραμμα COSME, ε, τη μεγάλη συνέργεια με το EIT, το Ινστιτούτο, αλλά θεωρούμε ότι ακόμα υπάρχει περιθώριο για να διευκρινίσουμε τις διάφορες πτυχές που αφορούν την πολιτική συνοχής. Ε, ε, αναφερθήκατε και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε ε, ότι μας ενδιαφέρει ε, και ήθελα να το θέξω διότι είναι ένα από τα θέματα που ανησυχούν περισσότερο τους συναδέλφους και το να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση προς αυτή την κατεύθυνση σίγουρα θα ενισχύσει την αριστεία και κατά συνέπεια όλο το ε, σύστημα έρευνας και καινοτομίας μας. Ένα δεύτερο ζήτημα και εσείς αναφερθήκατε σε αυτό όπως σας είπα, συμφωνούμε στη γενική τοποθέτηση του προγράμματος και συμφωνούμε ότι δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να υποστηρίζουμε και τη βασική έρευνα. Εσείς είπατε ότι δεν το λησμονούμε και το ξέρω γιατί σας γνωρίζω, αλλά ξέρετε πόσες φορές εμφανίζεται η έκφραση θεμελιώδης έρευνα στο επιστημονικό πρόγραμμα σε ένα έγγραφο 128 σελίδων. Ε, κάποιος με επεσήμανε ότι αναφέρεται μόνο δύο φορές. Πρέπει να πω ότι μας εξέπληξε αυτό και νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδιαφέρει ενδιαφέρει πολλούς από τους ερευνητές μας και τους ανησυχεί κιόλας. Και δεν θα πρέπει να ε, σας κρύψω ότι ανησυχούμε από πλευράς πολιτικής ομάδας για τα θέματα προϋπολογισμού, για τους διάφορους πυλώμενες και προγράμματα που περιλαμβάνει το Horizon 2020. Ένα παράδειγμα, ε, τα... Ε, ε κέντρα Marie Curie που ξέρετε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθά νέους ερευνητές να προχωρήσουν και να κινούνται στην Ευρώπη αλλά ο προπολογισμό που μας δίνεται είναι σίγουρα ανεπαρκής ε, προς το σημείο αυτό ιδίω δε αν το συγκρίνουμε με την προσαρμογή που προβλέπεται ε, για το EIT όπου ε, το έργο κατάρτισής του περιλαμβάνει πολύ, ε, έχει πολύ μικρότερες επιπτώσεις. Έχω πολλά ανησυχητικά στοιχεία για το EIT, αλλά βλέπω ότι με κοιτάει με το άγρυπνο βλέμμα της η πρόεδρος, μας δώσατε τα στοιχεία, θα τα συζητήσουμε, αλλά είναι πολλά τα χρήματα για το δεύτερο τμήμα, χωρίς το EIT, αντίθετα με το ERC, να αποτελεί τμήμα του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο θα μπορούσε να δώσει ίσως την εντύπωση ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας, το οποίο είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει και θα θέλαμε να ξέρουμε και την άποψή σας επ' αυτού. Και τέλος, ε, ε, έχω μεν και άλλα στοιχεία να σας πω, αλλά ε, επειδή θα πρέπει να ολοκληρώσω, κύριε Κουρέλ, μας είπατε ότι προχωρήσαμε πολύ τα θέματα της απλούστευσης, αλλά νομίζω ότι από αυτές τις συζητήσεις που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια, ήλπιζα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είχε φτάσει πολύ περισσότερο. Φαντάζομαι ότι ο συνάδελφος όμως θα εμβαθύνει περισσότερο από αυτού, επομένως θα σταματήσω εγώ εδώ σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριο Σέλλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε <clears throat> και αγαπητέ κύριε Γιάννη Σμιτ. Βέβαια σε πέντε λεφτά είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς και σαν σχιώδης εισηγητής και σαν συμμετέχον ευρωβουλευτής, αλλά θα προσπαθήσω να τα αναμίξω. Η πρώτη μου ερώτηση είναι σχετική με τον προϋπολογισμό. Οι αριθμοί φαίνονται καλή αύξηση κατά 49% αλλά πρέπει όλοι να γνωρίζουμε και εδώ στρέφομαι και προς το Κοινοβούλιο. Το 49% είναι καθαρά από τον προϋπολογισμό πρέπει δηλαδή ε, για να αντιπεξέλθουμε στον, στο, στην, ε, στον πληθωρισμό να αυξήσουμε ε, τον προϋπολογισμό κατά 15% μας μένει λοιπόν άλλο ένα 29% και βλέπουμε ότι έχουμε το EIT και το CIP οπότε συρρυκνώνεται ακόμη η αύξηση. Άλλωστε υπάρχουν διάφορα προγράμματα, προγράμματα που είναι ασαφή. Το ITER και αναφέρω και αυτό το οποίο δεν ανέφερε για τακτικούς λόγους Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το GMS, το οποίο όμως επίσης θα χρηματοδοτηθεί. Εάν λοιπόν σκεφτούμε και δεν θέλω εδώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες ότι είναι λογικό να μοιράζουμε την ίδια πίτα αλλά από την βασική έρευνα στην ουσιαστική ανάπτυξη και έρευνα ε, προς τις αποδείξεις και αν θέλουμε όλα αυτά να τα προχωρήσουμε μέχρι τους δημόσιους διαγωνισμούς για τα δημόσια έργα τότε ε, δεν υπάρχει τόση αύξηση του προϋπολογισμού. Και γι' αυτό τότε στρέφομαι προς τους Ευρωβουλευτές και ρωτώ, δεν αμφισβητώ εδώ τη θέση του ΕΛΚ ότι είχαμε αποφασίσει να διπλασιάσουμε τον προϋπολογισμό της έρευνας και είχαμε απαιτήσει 100 δις ε, ευρώ, διότι διαφορετικά θα διαπραγματευόμαστε για ένα πρόγραμμα πρόγραμμα όπου η κυρία Μαντουρέλ και άλλοι συνάδελφοι έχουν πολύ σωστές παρατηρήσεις για τα προγράμματα αλλά δεν ξέρουμε για ποιο όγκο μιλάμε. Εάν δεν επιτύχουμε τουλάχιστον τα 80 δις τότε εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούμε ε, να χρηματοδοτήσουμε ένα πρόγραμμα στο EIT ή ότι δεν θα χρειαστεί να διαγράψουμε ένα σωρό προγράμματα για να καλύψουμε άλλα τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε στο μέλλον. Θέλω λοιπόν καταρχήν να αναφερθώ στα προβλήματα ότι δεν είναι δυνατόν αν δεν έχουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο προϋπολογισμού να συζητάμε για συγκεκριμένα προγράμματα. Πιστεύω ότι η πρόταση είναι καλή, ότι η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου είναι καλύτερη παραποτέ. Ε, την στηρίζω και σαν εισηγητής και ε, τα έχω συζητήσει και σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους, αλλά είναι τα πρώτα σχόλια, η πρώτη αξιολόγηση, ε, πώς μπορούμε να προωθήσουμε τα πανεπιστήμια πώς είναι δυνατόν να προχωρήσουμε στα πλαίσια της πανεπιστημιακής έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και των συλλογικών οργάνων των εξωευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Γι' αυτό και είπατε πολύ σωστά ότι πρέπει να συνενώσουμε ε, για να μπορέσουμε ε, να συνδυάσουμε ε, την ε, χρηματοδότηση της, εξο, της εξωπανεπιστημιακής έρευνας στην Ευρώπη με την ενδοπανεπιστημιακή έρευνα. Και ε, όταν κοιτάξουμε τους κανόνες ε, συμμετοχής πώς θα συνεργαστούν η έρευνα και η καινοτομία διότι ένα Ινστιτούτο μπορεί να έχει ε, υποβάλει μία σωστή νομοθετικά πρόταση αλλά πώς αυτό θα μπορέσει να αξιολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εντάσσεται και στην καινοτόμα προσπάθεια. Είναι δηλαδή συγκεκριμένο συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε μεταξύ βασικής έρευνας, ε, απλής έρευνας, ε, προωθήσεως και πόσο θα διατυπώσουμε διάφορα μέτρα που να καλύπτουν όχι μόνο τις επιθυμίες μας αλλά και τις δυνατότητές μας. Και μία τελευταία ερώτηση προς τους ε, συνεργάτες μας, προς τους ε, ευρωβουλευτές. Πρέπει να συμφωνήσουμε για το τρίτο πρόγραμμα έρευνας ε, της Ευρώπης, ότι δεν θα διαχωρίσουμε στο EIT τις νομοθετικές εκθέσεις για τον ορίζοντα 2020, τους κανόνες συμμετοχής και τα υπόλοιπα θέματα, διότι έτσι απλώς θα αποδυναμώσουμε τη διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου. Πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε σοβαροί, να προχωρήσουμε δομημένα για να έχουμε μία πιο ισχυρή θέση διότι διαφορετικά μπορεί να ζητήσουμε πράγματα από τον ορίζοντα 2020 και επί της ουσίας να μην μας συμβουλευτούν καθόλου. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Ματίας έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω το λόγο στην Επιτροπή αυτή μετά την εκλογή σας. Θα ήθελα συνεπώς να σας συγχαρώ, να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία και ελπίζω να συνεχίσετε την εξαιρετική δουλειά ε, του ε, προκατόχου Προέδρου της Επιτροπής αυτής. Θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία. Δεν θα ήθελα όμω να αναφερθώ μόνο σε αυτό. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση. Αν έχει συγκεκριμένους στόχους στο Ινστιτούτο, ε, Βεβαίως ε, αυτοί οι στόχοι υποστηρίζουν το πρόγραμμα Horizon 2020. Αν όμως υπάρχουν και άλλα προγράμματα που υποστηρίζουν τους ίδιους στόχους, πρέπει να τα δούμε όλα μαζί ως σύνολο. Πρέπει λοιπόν ε, ως κοινοβούλιο, ναι με να εξετάσουμε τα διάφορα θέματα ξεχωριστά, αλλά να έχουμε μια κοινή θέση συνολική. Βλέπω με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις του Κοινοβουλίου, ειδικότερα όσον αφορά την απλοποίηση και πιστεύω ότι είναι πραγματικά μια μεγάλη πρόοδος αυτό ήδη. Όμω, θα ήθελα να δω και τις υπόλοιπες προτάσεις του Κοινοβουλίου να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το σύνολο ιδεών και ενιών που μας παρουσιάζεται εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε όμως στην αρχή μόνο μιας διαδικασίας και γι' αυτό Είμαι αισιόδοξη ότι θα έχουμε χρόνο να αναθεωρήσουμε, να εξετάσουμε εκ νέου ε, μερικές, ε, μερικές προτάσεις ε, και στο μέλλον. Θα ήθελα να επιμείνω σε ένα σημείο που μου φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, μια και βρισκόμαστε σε μια πρώτη συζήτηση σήμερα, δεν θα μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά κάτι το οποίο με ανησυχεί και πάντοτε με ανησυχούσε και μία ακόμη φορά το επαναλαμβάνω, συγγνώμη και ολα το επαναλαμβάνομαι, νομίζω ότι το πακέτο αυτό πρέπει να έχει μία ευρύτερη, έναν ευρύτερο προσανατολισμό, αλλά δεν θα πρέπει να είναι τόσο κλειστό όσο είναι τώρα, γιατί βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επιστήμη και η καινοτομία διέρχονται και αυτές κρίση και γι' αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα περιθώριο για έκτακτα προγράμματα που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας, Προκλήσεις που ενδεχομένως έχουμε ήδη εντοπίσει και ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες που δεν τις γνωρίζουμε ακόμα, μπορεί να μην τις είχαμε προβλέψει. Και γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να υπάρχει ένα τέτοιο είδους ε, περιθώριο για τα προβλήματα που θα προκύψουν στο μέλλον και που έχουν να κάνουν πράγματι με την κοινωνία. Είναι γεγονός ε, ότι η επιστήμη και η καινοτομία είναι τομείς ε, με ιδιαίτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και είναι ουσιώδους σημασίας για την ανάπτυξη των ικανοτήτων μας και ειδικότερα για την εξασφάλιση της ε, συνοχής μας ως Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γι' αυτό το λόγο λέω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, ο πλήρης διαχωρισμός ας πούμε, των στόχων ε, για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το πρόγραμμα Horizon 2020. Το έχουμε ξαναπεί αυτό σε πολλές συζητήσεις, υποθέτω ότι η συζήτηση θα συνεχίσει. Είναι προφανές ότι μιλάμε για ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προγραμμάτων με έναν συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ένα μόνο σενάριο, το σενάριο της συνοχής και χωρίς να συγχέουμε τους στόχους και το δικό μας ρόλο εδώ, στο συγκεκριμένο πακέτο του 2020, να μην αναφερόμαστε μεν να μην αναφερόμαστε μόνο σε, ένα, σε καθένα από τα προγράμματα αυτά μεμονωμένα. Πρέπει πάντοτε να βλέπουμε ευρύτερα το σύνολο των προγραμμάτων. Γιατί πρόκειται για στοιχεία που αποτελούν την ίδια την ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία ακόμη ανησυχία μου, ξέρω ότι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, γι' αυτό θα, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Η κυρία Μαντουρέλη ήδη αναφέρθηκε στο θέμα της ε, θεμελιώδους έρευνας. Δεν θα επιμείνω σε αυτό, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στις κοινωνικές επιστήμες. Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες είναι... Δεν πρέπει να, είναι, να θεωρούνται δεύτερης διαλογής ε, ε, πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα και αυτές. Είναι, είναι μια κοινή μας κληρονομιά. Και είναι κρίμα αυτή την κληρονομιά να μην τη χρησιμοποιούμε για να παρέμβουμε σε κοινωνίες που τις γνωρίζουμε καλά. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έχουν απλώς ένα συμβουλευτικό ρόλο στα επόμενα προγράμματα έρευνας και επιστήμης. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διαδοτικά ταμεία κυρίως για την ενίσχυση των ε, υποδομών προς αυτή την κατεύθυνση διότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος κάποιοι τομείς ε, της ε, έρευνας ε, να παραμείνουν ορφανές στην κοινωνία μας, για να το πω έτσι. Και αυτό βέβαια αποδυναμώνει και δεν ενισχύει τον Ευρωπαϊκό Χορό Έρευνας. Λοιπόν, επειδή πλατιάζω, θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινοτομίας και Τεχνολογίας συγκεκριμένα. Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση που γίνεται και που πρόκειται να γίνει. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία ήδη αναφέρατε εσείς στα εισαγωγικά σας σχόλια και στην παρουσίασή σας. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε, αλλά θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήματα πολύ συγκεκριμένα. Το πρώτο ερώτημα αφορά τον ορισμό των προτεραιοτήτων για τα κίξ γιατί νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ σαφέ και είναι μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε. Και το δεύτερο ερώτημά μου, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται μια περίοδο αναθεώρησης, είναι αυτό το accountability για το οποίο έχετε μιλήσει πολλές φορές. Δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, Συγγνώμη που μιλάω μόνο για τα προβλήματα και φαίνεται σαν να μην βρίσκω κανένα θετικό στοιχείο σε όλα τα μας είπατε. Ευχαριστώ κύριε Λάμπερτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ε, και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπρέτ ο οποίος έχει διευθύνει τις εργασίες εδώ και δυόμιση χρόνια. Δεν ε, θα ε, ασχοληθώ με την ουσία διότι δεν έχω εξετάσει τόσο ε, ακριβώς τον ορίζοντα 2020. Γι' αυτό θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τα βασικά σημεία εστίασης, επτά το σύνολο σε σχέση με το σύνολο, με το σύνολο του προγράμματος. Πρώτον, χρειάζεται καλή ισορροπία από τη θεμελιώδη έρευνα μέχρι την καινοτομία και νομίζω ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το έχουμε αυτό. Υπάρχει όμως ένας περιορισμός, δεν θέλουμε να πάμε πάρα πολύ μακριά όσον αφορά τις δραστηριότητες της αγοράς, γιατί είναι πέραν ε, του πεδίου εμβέλεια συγκεκριμένου προγράμματος. Δεν θέλουμε να επιδοτήσουμε ε, ε, τέτοιες δράσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως θα πηγαίνουν πολύ καλά. Διότι στο κάτω-κάτω της γραφής υπάρχει και ο ανταγωνισμός. Επίσης, πρέπει να υπάρξει μια ευθυγράμμιση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και χαίρομαι με το γεγονό ότι το πακέτο αυτό φαίνεται να ευθυγραμμίζεται πολύ περισσότερο με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα. Έχουμε και κάποιες ακόμα ανησυχίες που ανέφεραν και συνάδελφοι που πήραν το λόγο πριν από μένα όσον αφορά τη σχέση μεταξύ περιφερειακών και διαρθρωτικών ταμείων και αυτού του προγράμματος. Εκεί νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Αν θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε ε, την αποδοτικότητα της επένδυσης που θα κάνουμε, νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτή την εστίαση. Ναι, να μην περιορίσουμε πάρα πολύ το σύστημα, να μην το κάνουμε πολύ κλειστό. Συμφωνώ σε αυτό. Εστίαση όμω σημαίνει επιλογή. Και επιλογή σημαίνει ότι πρέπει να μείνουν ορισμένα πράγματα στι περιφέρειε στα κρατημέλη. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα πράγματα δεν θα ληφθούν υπόψη ή ότι δεν θα τα φροντίσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να αποφασίσουμε πού θα εστιάσουμε εμείς, πού θα ε, δοθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Κάτι ακόμη μεγαλύτερο περιθώριο για τους μικρότερους εταίρους, του μικρότερους παίκτε. Μικρότεροι εταίροι συχνά μα λένε ότι είναι πάρα πολύ δαπανηρό αυτό για μα, και γι' αυτό δεν συμμετέχουμε. Ξέρω ότι έχουν γίνει κάποια προσπάθεια όσον αφορά, κάποιες προσπάθειες όσον αφορά τους κανόνες ε, συμμετοχής τους. Ελπίζω να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε περαιτέρω αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά τώρα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρέπει η Ευρώπη να μπορεί να υποφεληθεί από τι δικέ τη δαπάνε και το λέω αυτό από στρατηγική απόψεω, αλλά από την άλλη θέλουμε και κανόνε πνευματική ιδιοκτησία, ε, τουλάχιστον ιδιοκτησία που προκύπτει από κοινοτικά κονδύλια. Θέλουμε αυτή η γνώση να κυκλοφορεί, να είναι μια ευκαιρία ε, δημιουργία αξίας, αλλά δεν θέλουμε αυτή η γνώση να μπει σε μια θηρίδα και να ε, είναι στα χέρια μεγάλων, λίγων και μεγάλων παικτών. Ένα πέμπτο σημείο που θα ήθελα να θέσω. Δεν θέλουμε αυτό το πρόγραμμα να είναι μια κρυμμένη πίσω πόρτα επιδοτήσεων ε, ή δώρων για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ξέρουμε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να ξοδέψουν χρήματα για την έρευνα και την ανάπτυξη. Θέλουμε να είναι καταλητικά αυτά τα κονδύλια σε σχέση με καινοτομίες που θα, ε, στις οποίες θα προβαίνουν κυρίως μικρότεροι παίκτες όσον αφορά τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ε, εμένα κάπως με ανησυχούσαν αυτές οι συνεργασίες Δεν ε, μας ενδιαφέρει πολύ το κόστος να, γίνεται, να κοινωνικοποιείται, αλλά το όφελος να ιδιωτικοποιείται. Το ίτερ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές και το περιθώριο που έχουμε για την επένδυση σε τέτοιου προγράμματα είναι ενδεχομένως ε, ε, ένα από τα τεράστια κομμάτια, τα οποία όμως αντλούν πάρα πολλούς πόρους. Και αυτό είναι κάτι που δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Αυτό το θέμα της χρηματοδότησης, της ε, στρατιωτικής τώρα έρευνας. Εγώ είμαι υπέρ της ε, ολοκληρωμένης άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι θα Ήμασταν πολύ καλύτερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση αν είχαμε κάτι τέτοιο από το να έχουμε 27 ξεχωριστές άμυνες, όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να ε, χρηματοδοτηθεί από εθνικούς προϋπολογισμούς. Και δεν θέλουμε από την πίσω πόρτα χρηματοδότηση για, εθνικές, ε, για εθνικούς μηχανισμούς άμυνας. Όχι, είναι αν αυτό δεν είναι μια κοινή ε, ευρωπαϊκή ε, αρμοδιότητα, εμείς πραγματικά είμαστε πάρα πολύ διστακτικοί. Αναφερθήκατε στα 80 δισεκατομμύρια, κύριε Έλερ. Δεν είναι και τόσα πολλά χρήματα αυτά, ώστε να έχουμε την πολυτέλεια να τα ε, διασπαθήσουμε στους διάφορους αμυντικούς μηχανισμούς των κρατών μελών. Λοιπόν, όσον αφορά τους κοινωνικούς επιστήμονες και την ασφάλεια, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα που υπόθηκαν σχετικά με αυτό το θέμα ε, είναι εντελώς άσχετα. Δηλαδή, αυτοί οι δύο τομείς δεν σχετίζονται μεταξύ τους και έτσι θα πρέπει να παραμείνουν άσχετος ο ένας με τον άλλον. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Έλερ για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Εγώ ήμουν τμήμα της συζήτησης για την ε, δέσμη 6 μέτρων, όταν συζητήσαμε και ήμασταν μια ενιαία ομάδα. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η προσέγγιση στην οποία αναφερθήκατε για το κατά πόσο εμεί συνεργαστήκαμε ω ε, εισηγητέ και σκιώδει εισηγητέ για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι θα επωφελούμασταν πραγματικά από μια ενιαία ολοκληρωμένη προσέγγιση και όχι να έχουμε ξεχωριστέ προσεγγίσει για ένα ε, κοινό θέμα. Ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο λοιπόν στον Γενικό Διευθυντή Ζαν Σμίτ για να δώσει ένα πρώτο γύρο απαντήσεων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θα κάνω απλώς γενικά σχόλια. Καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Μαντουρέλ, τον κύριο Έντελ, ε, Έλερ, την κυρία Ματίας και τον κύριο Λάμπερτς ε, για την ε, υποστήριξή τους και τα καλά τους λόγια για το πρόγραμμα. Ε, νομίζω ότι πολλά από αυτά επισημαίνουν ότι ακούσαμε τις προτάσεις σας στο παρελθόν και διαβάζουμε και τις εκθέσεις που μας υποβάλλατε. Υπάρχουν κάποια θέματα βέβαια τα οποία βαθύξατε. Καταρχάς, το κατά πόσο επαρκεί ο προπολογισμό. Νομίζω ο κύριος Έλερ αναφέρθηκε στο σημείο αυτό. Αυτό είναι βασικό σημείο βεβαίως και τα προγράμματα μεγάλης κλίμακας ε, έχουν μείνει εσκεμμένα εκτός αυτού του πακέτου, διότι αν πρέπει να απορροφηθούν και αυτά, σίγουρα δεν επαρκούν τα 80 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι σαφές. Αρκετοί αναφέρθηκαν στο θέμα της διεύρυνσης. Ε, ε, σας είπα ότι ε, είμαστε μια Ευρώπη των 27 κρατών μελών και η αριστεία υπάρχει παντού. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι αυτές οι πηγές αριστείας ε, θα βρουν χώρο να εκφραστούν στο Ορίζον 2020. Και γι' αυτό και πρέπει, και θα επανέλθω εδώ σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, να υπάρχει στενή σύνδεση με τα διαρθρωτικά ταμεία. Δεν θα πρέπει όμως να δημιουργηθεί μια κατάσταση στην οποία θα συγχέονται οι στόχοι. Όταν αναφερόμαστε στην ανάπτυξη ικανοτήτων σημαίνει ότι εξυγχρονίζουμε τα πανεπιστήμια, αγοράζουμε εξοπλισμό, ε, να βοηθήσουμε κάποιους επιτόπου να λάβουν επιδότηση και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για νέα διαρθρωτικά ε, ταμεία στο η νέα προγραμματική προγρα... κονδύλια από τα ταμεία συγγνώμη, στη νέα προγραμματική περίοδο που θα επικεντρωθούν ακριβώς στην έρευνα και στην καινοτομία εάν χρησιμοποιηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση, μπορούν να δημιουργήσουν δεξιότητες και ικανότητες ε, σε χώρους στους οποίους δεν υπάρχουν και σε χώρες τις οποίες δεν υπάρχουν. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει άριστη συμμετοχή στο Horizon 2020 και σε προηγούμενα προγράμματα. Έχουμε προγράμμα, ε, παραδείγματα. Η Ιρλανδία και η Ισπανία, για παράδειγμα. Χώρε που χρησιμοποιούν τα διορθωτικά ταμεία για να αναπτύξουν τι δυνατότητέ του στην έρευνα. Χρησιμοποιούν τα κονδύλια αυτά για να είναι βέβαιοι ότι έχουν μια καλή βάση γνώσεων και αυτέ οι χώρε συμμετέχουν πολύ καλά στο πρόγραμμα πλαίσιο. Αντίστοιχο παράδειγμα έχουμε και από την Πορτογαλία. Επομένω, θα πρέπει να δούμε τι σχέση υπάρχει μεταξύ διορθωτικών ταμείων και του ορίζοντα 2020 χωρίς να συγχαίουμε τα ταμεία. Νομίζω ότι η έκθεση του κυρίου Φανλίστερ αποτελεί πολύ καλό ε, τυφλοσούρτη για να μπορέσουμε να δούμε ε, τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Τώρα, οι βασικές προτεραιότητες, ε, οι ε, ηγετική θέση τη βιομηχανία και οι προκλήσει τη κοινωνία. Κάποιοι από εσά είπατε ότι δεν έχουμε επαρκή κονδύλια για τη βασική έρευνα, κάποιοι άλλοι είπαν ότι δεν έχουμε επαρκή κονδύλια για την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και κάποια άλλα φόρα μα είπαν ότι δεν έχουμε προ... κονδύλια για να αναπτύξουμε τι ε, προκλήσει τη κοινωνία. Αυτά βέβαια θα τα δούμε και σχετίζονται και με τα θέματα του προπολογισμού που ανέφεραν αρκετοί από εσά. Επαρκή απλούστευση έχει φτάσει μέχρι το σημείο που χρειάζεται. Ε, κατά την άποψή μας ναι, αλλά όταν φτάνουμε στην απλούστευση φτάνουμε απευθείας σε ένα πολύ πολύπλοκο ζήτημα και συζήτηση και είναι το εξή. Εμεί προτείναμε το ίδιο ποσοστό χρηματοδότηση για διάφορε φορολογικέ βάσει. Αλλά ορισμένοι λένε ότι το πανεπιστήμιο είναι διαφορετικό από μια μικρή επιχείρηση. Η μικρή επιχείρηση είναι διαφορετική από μια μεγάλη επιχείρηση. Το ερευνητικό Ινστιτούτο ε, είναι διαφορετικό από το ερευνητικό πανεπιστήμιο και το πανεπιστήμιο στο οποίο επικεντρωνόμαστε κυρίω στη διδασκαλία. Και εάν ξαναγυρίσουμε στο προηγούμενο, τι θα γίνει, ότι δεν έχουμε απλούστευση και πάλι. Και έχετε και τη δύσκολο έργο να το αποδείξετε σε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Εάν προσλαμβάνετε λιγότερου από όσου ε, προτείνει ο ορισμό για τη μικρομεσαία επιχείρηση, δεν έχετε χρηματοδότηση. Θα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν και να μην κάνουμε διάκριση μεταξύ του γιατί δεν έχουμε απλώστευση. Και εδώ φοβάμαι ότι πολλοί θα πούνε ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντε που συμμετέχουν και δεν μπορούμε να έχουμε ισότιμη μεταχείριση. Προσέξτε, σα εφιστώ την προσοχή, αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε απλούστευση. Αναφέρθηκαν και πάλι κοινωνικές επιστήμες. Δεν έχουμε πρόθεση να δώσουμε ζωτικό ρόλο στις κοινωνικές επιστήμες μόνο. Θέλουμε όμως να λάβουμε υπόψη και τους βασικούς παράγοντες για να αντιμετωπίσουμε τι βασικές προκλήσει τη κοινωνίας. Θέλουμε να βγουν από τον κλειστό τους ε, κύκλο, το, το συνεφάκι τους και να ε, μπορέσουν να δούνε τι γίνεται στην πραγματικότητα, είτε έχουμε τη γυράσκουσα κοινωνία ή την ασφάλεια. Ή μας ρώτησε η κυρία Ματίας τι σχέση έχει η ασφάλεια και με τις δύο έννοιες με τις προκλήσεις της κοινωνίας. Αν δείτε τα όσα συνέβησαν στο Λονδίνο πρόσφατα, δεν μπορείτε να μου πείτε ότι ασφάλεια και οι κοινωνικές προκλήσεις δεν έχουν καμία σχέση. Υπάρχουν ε, ε πηγές ε, τρομοκρατίας ε, και φονταμενταλισμού στις κοινωνίες μας και δυστυχώς δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει αυτά και για πολύ διάστημα τα έχουμε εκτός συζήτησης. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να τα συμπεριλάβουμε και αυτά στη συζήτηση. Ε, μια τελευταία ερώτηση για τους μικρούς ε, παίκτες. Όπως σας είπα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το πρόγραμμα Horizon 2020 ε, θα ε, επικεντρωθεί σε αυτούς, γι' αυτό λοιπόν έχουμε και χονδύλια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει και στα μικρά ερευνητικά πανεπιστήμια και Ινστιτούτα να συμμετέχουν. Ε, θα σταματήσω εδώ, ευχαριστώ την Επιτροπή σας για την υποστήριξη και επειδή και ο κύριος Ρόιλ ήρθε ε, μετά από την αρχική μου παρουσίαση, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την αγαστή συνεργασία στη διάρκεια της Προεδρίας του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομο γιατί αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξουν και άλλα ερωτήσει για την γενική προσέγγιση για το 2020. Ένα από τα βασικά θέματα είναι ότι καταρχήν είναι συμβατά με την προοπτική του 2020 και δεύτερον ότι έχουμε ορισμένα κριτήρια τα οποία παρουσιάζονται στην πρόταση και ε, έχουμε ορισμένα ορόσημα και άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και νομίζω ότι αυτά που έχουμε προτείνει είναι καλά και δεύτερον άπαξ και κατατίσουμε τα κριτήρια ο καθένας θα μπορέσει να καταλήξει τα συμπεράσματά του. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και πιστεύουμε ότι τα θέματα τα οποία προτείνουμε είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα προβλήματα της κοινωνίας και θα επανέλθω. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στον ισχύοντα κανονισμό και στα θέματα που εξετάσαμε στο τέλος ε, υπήρξε μια πολύ απότομη προσέγγιση, δεν υπήρχε μια βαθιά ανάλυση και πρέπει αυτή τη φορά να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε από καλύτερο σημείο. Ένα άλλο θέμα που έσθεσαν δύο βουλευτές είναι το θέμα της διαφανείας και του ε, απολογισμού και ε, υπάρχουν ε, κανονισμοί που αναφέρονται σε όλα τα γραφεία και που πρέπει να εφαρμόζουν τις αρχές το ανταγωνιστική της ανταγωνιστικής προσφοράς, της διαφάνειας κτλ. Και αυτό που είναι πολύ πιο σημαντικό είναι ότι ε, υπάρχει το θέμα της ε, απαλλαγής. Η EAT πρέπει άπαξ του έτους να έρχεται στο Κοινοβούλιο για να πάρει απαλλαγή και το Κοινοβούλιο έχει τον ίδιο ρόλο στην παρακολούθηση και στον έλεγχο των εξόδων του EIT όπως και οποιοδήποτε άλλου οργανισμού. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε. Το Ινστιτούτο είναι ευέλικτο και βεβαίως υπόκειται στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Γκλάντε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τους ομιλητές. Συμφωνώ με αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Θέλω όμως να τονίσω ε, για να επανέλθω στην ε, απάντηση του κυρίου Σμιτ σε θύματα του προπολογισμού. Ε, ξέρουμε τι γίνεται στο Κοινοβούλιο αλλά ξέρουμε τι γίνεται και στο Συμβούλιο και στα κράτη-μέλη και όλα αυτά πρέπει να τα εξετάσουμε στο πρόγραμμα πλαίσιο και να δούμε τι θα γίνει με τον ορίζοντα 2020 διότι το Φεβρουάριο θα έχουμε μία συνεδρίαση, ήδη καταρτήσει ένα ψήφισμα σχετικά. Πρέπει να εξηγιανθεί ο προϋπολογισμός αλλά δεν μπορούμε να εξοικονομούμε τα πάντα και για την ανάπτυξη. Ε, χρειάζεται και η έρευνα και ε, πρέπει να εξετάσουμε και από αυτήν την ε, ε, οπτική γωνία της εκθέσεις. Όσον αφορά σκιώδη, τη θέση μου σαν σκιώδη εισηγητή για αυτό το θέμα πρέπει να σας πω ότι ποτέ δεν έχω δει τόσες προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να γίνονται αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας συγχαίρω αλλά αντιλαμβάνομαι ότι πέραν αυτού πρέπει να υπάρχει ευελιξία και επίσης είναι καλό ότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί και ότι πλέον θα υπάρχει ένα συνομιλητής για πολλά θέματα. Και έχω τρεις ερωτήσεις. Καταρχήν, τι γίνεται για τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις σχετικά με ε, το πρόγραμμα COSMET. Δεύτερο, τι θα γίνει με τις συνεργασίες με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τρίτον το ε, γραφείο COST, τι ρόλο θα παίζει στο μέλλον Ευχαριστώ. Ο κύριος Φόρμπς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, η κυρία Φόρμς. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ρόιλι ε, για τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο υπερασπίστηκε το θέμα της αριστείας επί δυόμιση χρόνια και την κυρία Σαρτόνη η οποία απέδειξε ότι μπορεί να υπάρξει ε, μία ανισορροπία των φίλων χωρίς όμως ε, να ε, υπάρξει κίνδυνος για την αριστεία. Εδώ σε αφορά την μόχλευση των επενδύσεων για τις βιομηχανίες και τις μεγάλες και τις μικρομεσαίες ε, θέλω να αναφερθώ χωρίς να σχολιάσω τώρα τον προϋπολογισμό αλλά θέλω να σας πω ότι 80 δις είναι ένα τεράστιο ποσό και πρέπει να υπενθυμίσουμε στις χώρες μας σε όλους τους ερευνητές ότι τα χρήματα αυτά είναι πάρα πολλά και δεν τα συναντά κανείς καθημερινά. Πρόκειται για μια τεραστία επένδυση. Πρέπει λοιπόν αυτή η αρχή της αριστείας να υπερισχύσει και ε, να ε, στερεωθεί. Δηλαδή ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν από τους καλύτερους, από τους άριστους δεν θα πρέπει δηλαδή να αναδιοχετεύονται στους ίδιους οι οποίοι συμμετέχουν και στην, στον επόμενο διαγωνισμό οπότε πρέπει να συνεχίσουμε όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία θα ήθελα να πω ότι ένας άλλος μεγάλος κορβανάς χρησιμοποιείται στην έρευνα και τεχνολογία της γεωργίας δηλαδή όταν ασχολούμεθα με θέματα τροφή υγεία, ε, υγείας και ε, καλό θα είναι να δούμε πώς θα ευθυγραμμιστούν. Ε, συμφωνώ ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει απλώς μία απλοποίηση αλλά ότι θα είναι επί της ουσίας και πρέπει εδώ να αναφερθώ στους διαφόρους εμπλεκομένους αλλά και στις διάφορες μορφές της επιστήμης οι οποίες ενδέχεται να έχουν πιο υψηλό κόστος ε, αν χρειάζονται περισσότερες εργατόρες, είναι πιο περίπλοκες. Όταν λοιπόν προσιλωνόμαστε σε ένα ποσοστό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτή της μετακινήσεις και δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε ορισμένες έρευνες γιατί ενδέχεται αυτό να είναι μία άθελη ε, επίπτωση αυτής της προσπαθίας. Όσον αφορά λοιπόν την ισορροπία που επιζητούμε, εγώ δεν ε, ε, είμαι ε, μόνο εκπρόσωπος ομάδος μου, θα μιλήσω και προσωπικά. Οπότε θα ήθελα να συνεχίσω και να σας πω ότι στηρίζω τις διάφορες εκθέσεις που έχει καταρτήσει αυτή η Επιτροπή στο παρελθόν και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους συμμετέχοντες ότι <clears throat> θα πρέπει ναι με να υπάρχει κατανομή των πόρων αλλά θα πρέπει να καταβάλει κανείς ε, τα χρεστούμενα την κατάλληλη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχει και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβικής ε, διότι δεν ε, πρέπει να λέμε ότι ναι μεν αυτό προβλέπουν τα λογιστικά πρότυπα αλλά για πρακτικούς λόγους θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ε, θέλω να ε, επικροτήσω τις ε, ηθικές λύσεις στα κράτη-μέλη διότι πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή συνοχή και σχετικά με αυτό που είπαν οι συνάδελφοι σχετικά με την διαφάνεια του EIT το επικροτώ και το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ε, πολύ σημαντικό και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει ένα ε, ανταγωνιστικό ε, μια ανταγωνιστική στέρηση στην Ευρώπη σε σχέση με άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Η κυρία Μέρκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους κυρίους ορκυκλημένους ε, για την παρουσίασή τους. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Θα κάνω απλώς τις ε, ερωτήσεις μου, δεν θα πω τίποτε άλλο. Μιλήσατε, μιλήσατε για το πρόγραμμα Horizon 2020, αλλά μήπως μπορείτε να μας πείτε η Ένωση της Καινοτομίας και το Horizon 2020 τι διαφορά έχουν, τι θα παραμείνει από την ε, Ένωση της Καινοτομίας αν θα έχει ολοκληρωθεί πλέον ε, το Horizon 2020 γιατί μας ενδιαφέρει η απλούστευση όχι μόνο στα διαρθρωτικά ταμεία αλλά και στα γεωργικά ταμεία. Γι' αυτό ε, χαίρομαι ιδιαίτερος ε, με το σχόλιο που έκανε προηγουμένως η συνάδελφος Φόρντ. Αναφέρατε επίσης ε, τα ΚΙΚΣ, αλλά δεν άκουσα και πολλά για τις ε, συμφωνίες καινοτομία, οι οποίες κανονικά αντιμετωπίζουν και εκείνες τις κοινωνικές προκλήσεις. Υποτίθεται ότι τις ακολουθούν. Στην ε, Ένωση της Κοινοτομίας αναφερόμασταν ε, στο ότι θέλουμε να έχουμε ε, κάποιες, ε, να υπάρχει ανταπόκριση κοινωνικές προκλήσεις, αλλά λέγαμε να μην είναι πάρα πολλές, γιατί έξι είναι πολλές, και τελικά καταφέραμε να τις μειώσουμε σε τρεις. Όμως, Ίσως θα έπρεπε να τις επαραφέρνουμε τελικά στις έξι. Έχουμε τις κίξ, έχουμε τις κοινωνικές προκλήσεις, έχουμε τόσα πολλά πράγματα και δεν έχουμε ολοκληρώσει και με τα EIPs και παρόλα αυτά θα δρομολογηθούν κίξ το 2014, το 2017, ενδεχομένως και νωρίτερα. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε μια ευρύτερη θεώρηση, εν πάση περιπτώσει, όλων αυτών των εργαλείων, της πληθώρας εργαλείων ε, που ε, μας καταιγίζουν και ε, να δούμε και τι άλλους ε, θεσμούς έχουμε στη διάθεσή μας για να τα καταφέρουμε. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο αν είναι μικρό το ποσό που λαμβάνουμε θα είναι και μικρό το σύνολο όρων και προϋποθέσεων πρέπει να ισχύουν για να λάβουμε αυτό το ποσό. Νομίζω ότι και αυτό είναι σημαντικό. Μιλήσατε επίσης για την κοινωνική καινοτομία και μιλήσατε και για την προσοχή ε, στις ε, κοινωνικές και ανθρωπιστικές ε, επιστήμες. Βεβαίως η καινοτομία δεν είναι άμεσο αποτέλεσμα των κοινωνικών επιστημών, αλλά είναι ένας τρόπος ε, συνεργασίας. Οπότε πώς θέλετε να το επιτύχετε αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φανίστερ Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είστε νέα πρόεδρος και αναλαμβάνεται τα ενία αυτής της νέας πολιτικής. Χρειαζόμαστε κονδύλια και αν έχουμε λιγότερες επενδύσεις από τα κράτη-μέλη δεν μπορούμε να επιτύχουμε και πολλά πράγματα. Πώς λοιπόν ε, διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την περίπτωση. πώ ε, πώς τοποθετήστε μέσω μιας σύμβασης ε, εθνικής σύμπραξης. Διότι αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν μέσω συγχρηματοδότηση. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν πώ μπορούν να συμμετέχουν τα κράτη-μέλη σε αυτή τη σημαντική αύξηση. Από εκεί και πέρα. Συζητάτε το θέμα του κόστου. Ωραία, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο από αυτό. Και έχουμε και τα κέντρα ε, αριστεία. θα πρέπει να οργανώσουμε μια κοινή ακρόαση προκειμένου να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές, να έρθουν στο φως οι βέλτιστες πρακτικές. Θα ήθελα να πω ότι οι αρχικές μας θέσεις απέχουν κατά πολύ ε, και δεν νομίζω ότι μπορούμε να λάβουμε υπόψη ευθύ εξ αρχή την αριστεία και τους άλλου στόχου ε, τη συνοχή στην Ευρώπη και να του προάγουμε με τόσο διαφορετικέ απόψει υπάρχει το πρόγραμμα Region of Knowledge. Γιατί δεν ε, συμπεριλαμβάνονται τα προγράμματα αυτά ε, στα προγράμματα για να δημιουργήσουν και τοπικό ενδιαφέρον. Το EIT, όταν ξεκίνησε το EIT έπρεπε να είναι το βασικό στοιχείο. Ίσως είναι βέβαια ο πιο παραμελημένος γιος. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με αυτό. Ίσως να χρειάζεται να εντείνουμε περισσότερο τις προσπάθειές μας. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ε, πρώτα μια διακυβερνητική λύση και από εκεί και πέρα να περάσουμε στην ευρωπαϊκή λύση. Αυτή τη στιγμή πρέπει να επενδύσουμε σε περισσότερα σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε ίσως και να εξελιχθεί όπως πρέπει. Αλλά από ό,τι βλέπω έχει ήδη ε, κολλήσει τις πρώτες παιδικές ασθένειες και θα δημιουργηθούν προβλήματα. Ε, η κυρία Μέρκης αναφέρθηκε στον ηγετικό ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας. Κατ' εμέ αυτά θα πρέπει να είναι συνδυασμένα. Και αυτό βεβαίως ισχύει και για όλες τις παραγωγές και για όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι η βιομηχανία του μέλλοντος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Πώς θα διαχειριστούμε τα νέα προϊόντα, πώς θα διαχειριστούμε τις νέες παραγωγές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και πάλι ο λόγος λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ όλους τους εκπροσώπους για τις παρεμβάσεις τους. Αναφερθήκατε στην ποιότητα των κανόνων, με χαρά το ακούω αυτό. Αναφερθήκατε και στη σχέση μεταξύ δραστηριοτήτων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, μικρές επιχειρήσεις για το Horizon 2020 και το πρόγραμμα Κόσνερ. Το πρόγραμμα αυτό βέβαια δεν ασχολείται με την έρευνα και την καινοτομία, αφορά τις επιχειρήσεις και τα επιχειρηματικά μολύβα. Μοντέλα, εμείς ε, στο Horizon 2020 ασχολούμαστε με καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την έρευνα. Όσον αφορά τώρα την αριστεία, θεωρούμε ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να είναι ανταγωνιστική η Ευρώπη ε, με τον υπόλοιπο κόσμο. Με τη μετριότητα δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα και αυτό δεν ισχύει μόνο για την έρευνα, ισχύει και για το ποδόσφαιρο και ισχύει και για τα πάντα. Μπορούμε να κερδίσουμε τον υπόλοιπο κόσμο μόνο μέσω της αριστείας, γι' αυτό και η αριστεία θα είναι το βασικό κριτήριο, βεβαίως μαζί με τις επιπτώσεις, αλλά είναι πολύ σημαντικά τα κριτήρια αυτά για τα προγράμματα. Όπως είπατε και εσείς αναφέρθηκαν και άλλοι στη σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία και η ιδέα του κυρίου θέλει να οργανώσουμε μια κοινή ακρόαση ίσως θα είναι καλή, διότι πολύ συχνά αναφερόμαστε ο ένας τον άλλον, αλλά καλό θα ήταν να μιλήσουμε από κοινού οι αρμόδιες επιτροπές. Ε, ναι, άκουσα, υπάρχει απλούστευση, αλλά υπάρχουν διάφορε μορφέ έρευνε. Ένα πράγμα έχω μάθει εγώ. Υπάρχει καλή και κακή έρευνα και δεν μα ενδιαφέρει η εφαρμοσμένη ή θεμελιώδη έρευνα. Ε, όσον αφορά την έρευνα, λοιπόν, θα πρέπει να κοιτάμε ο ένα τον άλλον στα μάτια και να δούμε αν θέλουμε να προχωρήσουμε ή να έχουμε όλε αυτέ τι παρεκκλήσει για την τάδε ή τη δίνα μορφή έρευνα. Και επίση, επαναλαμβάνω πόσο σημαντικέ είναι και πάλι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει για το θέμα αυτό. Η κυρία Μάρκη ρώτησε τώρα τι σχέση υπάρχει μεταξύ του ορίζοντα 2020 και τη καινοτομία και την Ένωση Καινοτομία. Για μα, η Ένωση τη Καινοτομία ήταν μια δέσμη μέτρων για να ενισχύσουμε το κλίμα τη καινοτομία στην Ευρώπη. Ε, μια δέσμη μέτρων που περιλαμβάνε 14 μέτρα για την πιο ευφυή χρήση των ε, μειοδοτικών διαγωνισμών και των δημοσίων προμηθειών, ε, μεταφορά τεχνογνωσίας, η οποία θα μπορούσε να είναι καλύτερα, ε, καλύτερα συστήματα διδακτορικών διπλωμάτων, ώστε να υπάρχει και ένα τμήμα ε, εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης στο βιομηχανικό κλάδο. Ε, Χρειάζονται λοιπόν πολλά μέτρα για να βελτιωθεί το κλίμα της καινοτομίας στην Ευρώπη και τμήμα αυτών είναι ο μηχανισμός χρηματοδότησης για τον ορίζοντα 2020. Το ορίζον 2020 δηλαδή είναι τμήμα της, Ένωσης, της εφαρμογής της Ένωσης Καινοτομίας, αλλά αν θέλουμε να έχουμε μια Ευρώπη καινοτομίας και θέλουμε η Ένωση Καινοτομίας να είναι η Ευρώπη της καινοτομίας, θα πρέπει να γίνουν πολλά στον τομέα της νομοθεσίας, ώστε να μπορέσει ο επιχειρηματικός κλάδος, ε, να μπορούν οι επιχειρήσεις να συστήνουν γίνονται πολύ γρήγορα και πολλά από αυτά τα μέτρα πρέπει να ληφθούν σε εθνικό και όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ρωτήσατε επίσης ε, ποια η σχέση με τις συμπράξεις καινοτομία οι συμπράξεις καινοτομία δεν είναι μέσο, είναι φόρα τα οποία ε, συγκεντρώνουν διαφόρους ε, ε, τομείς της κοινωνίας για να συζητήσουν τα διάφορα θέματα. Αν δείτε για παράδειγμα το θέμα της ενεργού γύρανσης, αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει να διαμορφωθεί η ερευνητική ατζέντα για τον τομέα της υγείας του ορίζοντα 2020. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συμπράξεις καινοτομία και να προχωρήσουν οι δραστηριότητες που βλέπουμε για τις προκλήσεις αυτές. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, προκλήσεις στην κοινωνία. Μακάρι να μπορούσαμε να αρκεστούμε στις έξι αυτές που έχουμε. Ε, μέχρι να ολοκληρώσουμε με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα είναι περισσότερες από έξι. Εάν μπορέσουμε να τις περιορίσουμε στις τρεις είμαστε πολύ ανοιχτοί για συζήτηση γιατί είναι πολύ σημαντικό να καθορίσουμε προτεραιότητες και αν μπορέσουμε να περιορίσουμε τον αριθμό των προτεραιοτήτων και τον αριθμό των μέσων ακόμα και μετά από τη μακρά και έντονη συζήτηση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου θα είναι επίτευγμα. Οι έξι λοιπόν λοιπόν, εάν μπορέσουμε να το περιορίσουμε στους έξι μόνο, θα είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα. Κοινωνική καινοτομία, έχετε δίκιο, αυτό δεν έχει σχέση μόνο με την τεχνολογία, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες δράσεις και νομίζω ότι αυτό είναι νέο στοιχείο για μας η κοινωνική καινοτομία. Δεν έχουμε κάνει πολλά στον τομέα αυτό. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι πολλά από τα καινοτόμα στοιχεία δεν προέρχονται από την τεχνολογία, προέρχονται από νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέο τρόπο δραστηριότητας. Είναι κάτι λοιπόν νέο και σίγουρα θα ξεκινήσουμε με πιλωτικά προγράμματα πριν περάσουμε σε μεγάλης κλίμακας προγράμματα. Ο κύριος Ρόι αναφέρθηκε και πάλι ε, στη σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία, αναφερθήκατε στην ακρόαση και νομίζω ότι όταν, ε, όπως και η κυρία Φόρντ, λέτε και εσείς ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι σημαντικές, αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι υπάρχουν και πολλές μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη που ακόμα αποσχολούν εκατομμύρια ανθρώπων και θα θέλαμε να παραμείνουν αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό. Στο 7ο πρόγραμμα ε, πλαίσιο έχουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ε, συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα και χρήση των διαθροτικών τομέα και θέλουμε να συνεχιστεί αυτό γιατί θέλουμε να έχουμε αυτή τη μεγάλη βάση στην Ευρώπη. Ναι, πρέπει να επικεντρωθούμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις μεγάλες επιχειρήσεις γιατί είναι πολύ σημαντικές για την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ευχαριστώ κύριος Κάτι ακόμη θα ήθελα να πω σε σχέση με το EIP, το, με το το, τα KICS κλπ. Ο συντονισμός όλων αυτών των πρωτοβουλίων είναι πολύ σημαντικός ε, γιατί όντως υπάρχουν διάφορες οπτικές γωνίες για να ειδωθούν όλα αυτά και με διαφορετικό τρόπο. Είναι σημαντικό είναι να έχουμε την ευρύτερη εικόνα όπως επίσης και να εξεύρουμε μηχανισμούς ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη σε σχέση με τα αποτελέσματα και να είναι ε, να διαδίδονται σωστά τα αποτελέσματα αυτά. Όσον αφορά τώρα τα, την ε, βιομηχανία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν και οι μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό η συμμετοχή αυτή της βιομηχανίε. Και νομίζω ότι είναι και κάτι το πολύ ενθαρρυντικό. Κάτι το οποίο είπε και ο κύριο Ροϊ, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι για τα αποτελέσματα. Έχετε απολύτω δίκιο. Πρέπει να εστιάσουμε στα αποτελέσματα και ειδικότερα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία. Έχουμε κάποια αποτελέσματα, ξέρουμε τα αποτελέσματα των ΚΙΚΣ, έχουμε κάποια απτά αποτελέσματα σε σχέση με τι νεοσύστατε επιχειρήσει, ε, με την ε, κατάρτιση ορισμένων ε, φοιτητών σε πανεπιστήμια που συμμετείχαν στα ΚΙΚΣ Όμω, όμως επειδή τα Geeks ε, υπάρχουν εδώ και 1,5 χρόνο μόνο, ε, δεν έχουμε παραπάνω αποτελέσματα. Κάποια όμως υπάρχουν και ευχαριστώ να τα μοιραστούμε μαζί σας, τα αυτά αποτελέσματα και με τον τρόπο μάλιστα που προτιμάτε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Όπως γνωρίζετε, σήμερα έχουμε και την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατόπιν θα υπάρξει ένα δεύτερο στάδιο πρώτη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μα. Έχω ένα μακροσκελέστατο κατάλογο εδώ και θα ήθελα να προτείνω στους συναδέλφους που θα λάβουν το λόγο τώρα να μιλήσουν για ένα-ενάμιση λεπτό για να θέσουν την ερώτησή τους, ώστε να υπάρχει χρόνος να σας δώσουν απάντηση οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από εκεί και πέρα να απαντήσουν και οι ε, Ευχαριστώ. <clears throat> Η πρόταση της Επιτροπής είναι πολύ καλή αλλά υπάρχουν ορισμένα θέματα που μπορούν να βελτιωθούν. Και ξεκινώ. Το περιεχόμενο είναι ισοσκελισμένο. Πολύ σωστά είπαστε ότι χρειάζεται και αριστεία και επέκταση, αλλά πρέπει τα δύο θέματα να είναι συμπληρωματικά, να υπάρχει κάποια συνέργεια μεταξύ των διαφόρων τρόπων ε, χρηματοδοτήσεως και όπως είπε και ο κύριος Βανλίσης Ρόι πρέπει να βελτιώσουμε την ε, περιφέρεια γνώσης. Ε, υπάρχουν και άλλα θέματα στον τομέα της αριστείας αλλά πιστεύω ότι μπορείτε να προχωρήσετε και περαιτέρω. Και να αναφερθείτε και στις ε, κοινωνικές προκλήσεις ε, και να δημιουργήσετε, ε, να απαντήσετε σε νέες προκλήσεις ενώ εσείς είπατε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες προκλήσεις. Επιπλέον πρέπει να πούμε ότι εδώ είναι ο κατάλληλος χώρος όπου οι μεγάλες βιομηχανίες μπορούν να συνεργαστούν με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πρέπει να βρεθεί η δυνατότητα να συνεργαστούν. Όσον αφορά τις κοινωνικές επιστήμες, θα πρέπει να υπάρξει ευελιξία και να υπάρχει μία πολυσχηδής προσέγγιση. Όσον αφορά τον ορίζοντα 2020 ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν δομικό συστατικό για να αντεπεξέλθουμε του κατακαιρματισμού και να προχωρήσουμε σε βασικούς τομείς όπως ο τομέας της ερεύνης για την υγεία στην Ευρώπη. Και τέλος όσον αφορά την απολοποίηση. Είμαι πολύ ευτυχής για τις προτάσεις τις οποίες έχετε υποβάλει και πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσουμε το ΦΠΑ και να στηρίξουμε το ΦΠΑ στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Πρέπει να δούμε τα ποσοστά, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι κάποιος τρόπος κατά αυτόν τον τρόπο να χρηματοδοτούμε την προστιθέμενη αξία και να απασχολούμε τους νέους ερευνητές. Αλλά βλέπω τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν σε ορισμένους ερευνητές και θα πρέπει ε, να βρούμε ένα γενικό κανόνα ο οποίος θα ισχύσει και κάτι διαφορετικό για την έρευνα για να υπάρχει σωστή χρηματοδότηση. Έχω και άλλες πολλές παρατηρήσεις αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Ναι, αλλά έτσι δεν επιτρέπεται στους υπολείπους να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Πρόντι. πολύ γρήγορα. Αφήνω όλους τους προλόγους. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε ενώπιον μίας ανάγκης να ξεφύγει ο πολιτισμός μας από την ύλη, ε, τουλάχιστον μερικός για να περάσουμε στο εγχώριο ακαθάριστο προϊόν. Πρέπει να καταλάβουμε πόσο κεντρικό ρόλο έχει ο άνθρωπος και πόσο σημαντικές επιπτώσεις έχουν οι δράσεις μας στη βιωσιμότητα. Γι' αυτό ακριβώς οι συνέπειες θα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει σύγκληση μεταξύ των ανθρωπιστικών σπουδών και των επιστημονικών σπουδών. Θα πρέπει να ξέρουμε τι άνθρωπο θέλουμε να προάγουμε και πώς μπορούμε να εξεύρουμε τη δέουσα ισορροπία με τη φύση και τον κόσμο. Να χρησιμοποιούμε με ευφυή τρόπο κοινά υλικά όπως για παράδειγμα ο γραφίτης και θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω και την ανάγκη να υπάρχει σύγκληση για την ανησυχία για την σωματική και πνευματική υγεία, διότι πολύ συχνά εξετάζονται ξεχωριστά. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι υπάρχει ένα μέσο το οποίο έχει στη διάθεσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ΣΤΟΑ, η οποία φυσικά είναι στη διάθεσή σας για να εμβαθύνουμε και αυτές τις πτυχές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πρόντι, η κυρία Τόγια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πρώτη παρατήρηση, πέρα από το γεγονό ότι εκτιμώ τα πολλά θετικά στοιχεία τα οποία είχε προτείνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έγιναν δεκτά, η πρώτη μου λοιπόν παρατήρηση είναι ότι εκτιμούμε ότι υπήρχε και μεγαλύτερο συντονισμό σε αυτή την προσπάθεια μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι το οποίο δεν είχαμε διαπιστώσει στο παρελθόν και ήταν ένα από του γόρδιου δεσμού ε, των προβλημάτων που αντιμετωπίζαμε. Ελπίζω λοιπόν να συνεχίσετε προ αυτή την άγουσα και να είναι διαρθρωτική αυτή η αλλαγή. Τι έγινε με την πτυχή του πολιτισμού, κάτι ακούστηκε, αλλά ε, ε, το λέω όχι γιατί μόνο η χώρα μου ακολουθεί το πρόγραμμα Cultural Edifice, αλλά γιατί ο πολιτισμός είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο πολλών ευρωπαϊκών χωρών και ως βιομηχανικό προϊόν. Ακούσατε την ομάδα υψηλού επίπεδου του οποίου ηγείται ο καθηγητής, του οποίου μου διαφεύγει το όνομα, που έχει έρθει επανειλημμένος εδώ στην Επιτροπή μας και είπε πόσο ενδιαφέρον θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία με καινοτρόμο τρόπο. Πρόκειται για κάτι το οποίο ετοιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είδαμε το υλικό. Ε, προσκόμματα τώρα στην πρόσβηση. Πολλέ φορέ ο πανεπιστημιακό κόσμο, ο κόσμο των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων δεν συμμετέχει γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, αντέξουν το κόστο του προγραμματισμού επειδή είναι αβέβαιο το κατά πόσον από εκεί και πέρα θα λάβουν τη χρηματοδότηση. Πολύ καλά να έχουμε νέα μέσα χρηματοδότηση, Αυτή τη στιγμή κάποιο έχει κερδίσει το μειοδοτικό διαγωνισμό και έχει λάβει τη χρηματοδότηση. Αλλά πώ μπορεί κάποιο ε, να επενδύσει χωρί να σπαταλεί τα χρήματά του. Ο προγραμματισμό είναι σημαντικός για να αυξηθεί ο αριθμό αυτών που έχουν πρόσβαση. Με την ελπίδα από εκεί και πέρα ότι θα έχουμε έρευνα και καινοτομία γιατί όσε περισσότερες πόρτες ανοίγουμε τόσα περισσότερα ανακαλύπτουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κέλλη. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να διαφωνήσω με τη γενική τάση και την ουσία αυτής της ε, προσπάθειας. Προφανώ είναι ευκταία όλα αυτά που μας λέτε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη συζήτηση που έχουμε σήμερα το βράδυ αλλά υπάρχουν ζητήματα όπως η απλοποίηση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα να ακούσω λίγο περισσότερα για αυτό το θέμα, ενδεχομένως όχι σήμερα. Και το θέμα που έθεσε ο κύριος Σμιτ σε σχέση με την προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων ερευνητικών ταλέντων στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ε, σε σχέση τώρα με τη χρηματοδότηση, νομίζω ότι λόγω της στρατηγικής 2020, λόγω της οικονομικής κρίσης, η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται ε, με κλάδους που μπορεί να αποδώσουν. Νομίζω ότι αναφέρθηκε στο ότι είμαστε, έχουμε μανία με τους ελέγχους. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μανία για τα επόμενα χρόνια με τη ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ε, με την αποδοτικότητα. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τεθούν στο περιθώριο μέχρι να έχουμε θέσεις απασχόλησης και ανταγωνιστικότητα που θα επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα στην Ευρώπη. Ε, αν λοιπόν θέλουν κάποιοι να ερευνήσουν, να μπορούν μπορούν ε, να έχουν πρόσβαση σε κονδύλια. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι για τα επόμενα 7-8 χρόνια ε, πρέπει να μπορούν να ε, δουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης να επιστρέφουν στην Ευρώπη. Κύριε Δελκαστήγιο, ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό τον πολύ γρήγορο κατάλογο παρατηρήσεων που έχουμε θα μπορέπει να γίνουν πολύ περισσότερα και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γενικό Διευθυντή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν γέννη για την προσπάθεια που έκαναν και τη δυνατότητα που έδωσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να συνεισφέρει, το οποίο βλέπουμε ε, ότι έχει ληφθεί και υπόψη και συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις μας ε, στην πρότασή σας. Θα σταθώ επιγραμματικά σε κάποια ε, στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Ε, υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία θα θέλαμε να συζητήσουμε από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα θέλαμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο επιτέλους να τα δούμε και στο τελικό έγγραφο το οποίο θα εγκρίθηκε στην Ολομέλεια. Υπάρχει περιθώριο για πολλά πράγματα, παρά το γεγονός ότι εγώ συμφωνώ με τα πιο ισιώδη στοιχεία αυτής της πρότασης και με τη δομή που έχει ε, χρησιμοποιηθεί και με το γεγονός ότι υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση υπό την ε, σκέπη του τριγώνου της γνώσης. Υπάρχουν όμως κάποια σημεία τα οποία με ανησυχούν. Ε, καταρχάς ε, είπατε ότι δεν είναι σαφής η σχέση και η συνέργεια με την πολιτική συνοχής. Αναφερθήκαμε στις περιφέρειες της γνώσης, αλλά χάθηκαν ε, και τα research potential εντό εισαγωγικών. Και αυτό είναι κρίμα, διότι... Ε, τα θέ, οι στόχοι της αριστείας και της συνοχής είναι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πολύ διαφορετικά μεταξύ των. Θα ήθελα να αφαιρθώ και στον προϋπολογισμό, πέραν του γενικότερου προβλήματος που έχουμε, για το ποιος θα είναι τέλος ο, επιτέλους ο προϋπολογισμός, ε, Κυρίως ε, με ενδιαφέρει το θέμα των υποδομών. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει ε, μεγάλο τμήμα του προϋπολογισμού το οποίο να είναι αφαιριωμένο στις υποδομές όπως ε, γίνεται και με το πρόγραμμα Marie Curie που έχει πάρα πολύ σημαντική προστιθέμενη αξία και είναι κρίμα που δεν αυξήθηκε επαρκώς ο προϋπολογισμός του. Και τέλος, μου έλεγε ένας ερευνητής πρόσφατα ότι φαίνεται ότι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η απλούστευση είναι ένας τρόπος να μειωθούν τα σφάλματα. Ενώ στην πραγματικότητα η απλούστευση θα πρέπει να είναι ένα μέσο ώστε ο συμμετέχον ή οι συμμετέχοντες να έχουν περισσότερες δυνατότητες. Και προς αυτή την κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει τεράστια προσπάθεια, ακόμα έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Πρέπει να συμβουλευτούν κάποια σημαντικά στοιχεία. Ε, η αμοιβή ανάλογα με το έργο που υλοποιήθηκε, για παράδειγμα, στις διάφορες ε, κοινοπραξίες. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ και πάλι όλους τους ε, ευρωβουλευτές οι οποίοι ε, παρέμβησαν διότι ε, όλοι τόνισαν την σημασία της σχέσεως του ορίζοντα 2020 και άλλων προγραμμάτων. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη στο ΦΕΤΣ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς και επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε με τις μεγάλες βιομηχανίες όπως είπε η κυρία Φόρτ και ο κύριος Βανίστελ Ρόι. Απλοποίηση. Χαίρομαι διότι εσείς έχετε εφαρμόσει την αρχή απλοποίησεως και ε, εντοπίσατε το βασικό θέμα, το θέμα ε, του πλήρους κόστους ενώ απλοποίηση σημαίνει ότι οι ε, κανόνες πρέπει να είναι πιο απλοί και εναρμονισμένη και να αποφύγουμε να έχουμε πάρα πολλούς χαμένους διότι δεν πρέπει ε, να χάσουμε ε, σε σχέση με άλλα προγράμματα. Ε, βεβαίως αναφέρθηκε το θέμα της αποτελεσματικότητας των πόρων που είναι πολύ σημαντικό το θέμα του συσχετισμού της φυσικής και της πνευματικής υγείας. Είδατε ότι ότι υπάρχει στενή σχέση και η κυρία Τόγια αναφέρθηκε στο, στην πολιτιστική κληρονομιά αλλά και στα διαρθρωτικά ταμεία, πράγμα που είναι σημαντικό για, για να μπορέσει κανείς να απαντήσει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Είπατε ότι χρειάζεται μια ομάδα υψηλού επίπεδου που να ασχολείται με τις τεχνολογίες, παρακολουθούμε την Επιτροπή αυτή, ακούμε τι έχουν να μας πούν και τον τονίζουν ότι πρώτα πρέπει να αναπτυχθεί η Ευρώπη. Η σύστασή τους είναι η έρευνα να χρησιμοποιηθεί καταρχήν στην Ευρώπη και εμείς αποφασίσαμε να μην το χρησιμοποιήσουμε για εύλογους ε, λόγους και είναι ένα θέμα που ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω. Επίσης με τις ε, απλοποιήσεις προσπαθήσαμε να καταργήσουμε τα εμπόδια κατά τρόπον ώστε οι μικρές επιχειρήσεις, τα μικρά ερευνητικά κέντρα να μπορούν ε, να έχουν πρόσβαση στα προγράμματά μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, ανάπτυξη για την οικονομία μας αυτό είναι το ρεφρέν του προγράμματός μας και γι' αυτό και σας είπα ότι για να προχωρήσουμε χρειαζόμαστε ε, ανάπτυξη διότι δεν μπορούμε απλώς με την λιτότητα και την πειθαρχία να προωθήσουμε την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε και αναπτυξιακά μέτρα. Και τέλος η κυρία Καστήλιο σχετικά με την ασύνδεση με τα διαρθρωτικά ταμεία είπατε ότι έπρεπε έπρεπε να έχουμε κάνει περισσότερο για τις υποδομές της ερεύνης αλλά βλέπετε ότι ε, δεν χτίζει κανείς μόνο με τα τούβλα και ε, ε, το, τα δομικά υλικά αλλά θα πρέπει να υπάρχει διασύνδεση και γι' αυτό εμείς έχουμε υπόψη μας και το πρόγραμμα μαρί και θα μπορέσουμε να επιτρέψουμε ε, πλήρη κινητικότητα όχι μόνο στο ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά και στο πρακτικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τρία λεπτά στη διάθεσή μας. Έχουμε τρεις εισηγητές ε, παρόντες. Εάν δώσουμε λοιπόν ένα λεπτό στον καθένα, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ξαναγίνει η συζήτηση και θα έχουμε και άλλα ανταλλαγή απόψεων, να δώσω λοιπόν καταρχάς το λόγο στην κυρία Ρέιρα Μαντουρέλ. Θέλετε να πείτε κάτι? Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Εγώ σημείωσα ε, πολλές πληροφορίες οι οποίες θα μου είναι χρήσιμες για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε στη συνέχεια, τι θα συζητήσουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία ετέθησαν εκεί, εδώ. Δεν θα πω περισσότερα, έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ τους ε, δύο διευθυντές που ήταν παρόντες εδώ και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σέλερ.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 Κύριε Σμιθ, πολλοί σας επένεσαν σήμερα, αλλά τώρα στα γρήγορα ε, θα αναφέρω κάποια προβλήματα. Το EIT είναι ε, το, ο πρώτος τάφος των φαραώ του 21ου αιώνα που περιέγραψε ο κύριος Μπαρόζο και δεν θα το στηρίξουμε. Το Risk Sharing Facility θα πρέπει να γίνει πιο ουσιαστικό για την πρόθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αποφυγή των μεσαζόντων. Θέλουμε να ξέρουμε τι, πώς θα χρησιμοποιήσει τους πόρους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι εννοεί. Θα θέλαμε ένα αυτούσιο πρόγραμμα έρευνας γιατί ήταν συμβιβαστική η λύση να το ενσωματώσουμε κάπου αλλού και θα πρέπει να είναι αυτούσιο γιατί έχει άλλους κανόνες. Εμείς δεν μιλάμε μιλάμε για στρατιωτική έρευνα αλλά έρευνα ασφαλείας και τέλος πρέπει από κοινού να δούμε πώς θα συνδυάσουμε τον ορίζοντα 2020 με τα διαρθρωτικά ταμεία διότι διαφορετικά δεν θα προχωρήσουμε. Πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η γέφυρα μεταξύ των δύο διότι διαφορετικά δεν θα έχουμε τη χρηματοδότηση για την αναγκαία καινοτομία στην Ευρώπη και θέλουμε μία συγκεκριμένη πρόταση για το πώς θα επιδράσουν τα δύο αυτά προγράμματα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να επαναλάβω σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Σμιτ ε, στην προηγούμενη του παρέμβαση, δηλαδή ότι θα υπάρξουν ε, μέτρα ανάπτυξη και όχι μόνο μέτρα λιτότητα. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πώ θα χρησιμοποιήσουμε το δημόσιο χρήμα, γιατί δημόσιο χρήμα θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση τη καινοτομία, τη έρευνα και πρέπει να δούμε κατά πόσο θα είναι τα αποτελέσματα ε, τα επιθυμητά ή όχι. Δεν πρέπει να ευνοούμε μόνο τις ε, προτάσεις ε, που αφορούν το τελικό προϊόν, γιατί μερικές φορές τα προϊόντα αυτά δεν ενισχύουν την ανάπτυξη, αλλά ενισχύουν τις ανισότητες που ήδη υπάρχουν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό τμήμα της, των μελλοντικών μας συζητήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ματίας. Ευχαριστούμε τους ε, διευθυντές ε, πέρα στις συνεδρίασεις για σήμερα. Αύριο το πρωί θα έχουμε συνεδρίαση των συντονιστών στις 9.30 και επομένως η συνεδρίαση της Επιτροπής θα συνεχιστεί στις 10.30 αύριο. Ευχαριστώ πολύ όλους. Καλό βράδυ. Η Πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς και ζητά συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση.